Iniziamo. Benvenuti a tutti. Σας καλωσορίζω όλους. Αρχίζουμε σας παρακαλώ με τις εργασίες της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, καταρχήν ε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σήμερα υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Γεωργίας, θα διοργανώσει μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη γεωργία. Γεωργία, ένα επικίνδυνο επάγγελμα. Πώς να βελτιώσουμε την υγεία και την ασφάλεια. Η κοινή αυτή ακρόαση με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνει στις 20 Μαρτίου του 2013. Εξάλλου η σημερινή μας συνεδρίαση όπως γνωρίζετε μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Μπορούμε να αρχίσουμε το σημείο 3, παρουσίαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, μίας μελέτης σχετικά με τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χέρμαν Φοντιέ, που είναι ο επικεφαλής της αρχής αυτής, της μονάδας, και θα μας μιλήσει για τους κινδύνους ε, από αυτά, αυτών των λοιπασμάτων Και αν και Των εντομοκτώνων, με συγχωρείτε. Στη συνέχεια, με την παρουσίαση του κυρίου ε, Μπορς, του Επιτρόπου, θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα και πρωτοβουλίες σε σχέση με την υγεία και προστασία των καταναλωτών. Ζωζε Μποβέ. Μία ανακοίνωση έλαβα ε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από έναν υπεύθυνο του, της Swedish Match που είναι μια σουηδική εταιρεία καπνών και που αναφέρει ότι η οδηγία περί καπνού θα συζητηθεί με την, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής Γεωργίας. Ως προς αυτή την πρόσκληση της Swedish Match, έγραψα στο Κοινοβούλιο και στους Προέδρους των Επιτροπών, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνάντησης με τους εκπροσώπους των εταιριών καπνών, διότι η δυνάμη του άρθρου 5.3 του κανονισμού περί υγείας ορίζονται οι όροι συνάντησης και τόνισα ότι θα συναντηθώ με τα πρόσωπα αυτά όταν συσταθεί το κατάλληλο πλαίσιο, διότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με την καπνοβιομηχανία. Δεν ξέρω εάν λάβατε την ίδια πρόσκληση, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ε, σαφείς και να υπάρχει διαφάνεια, διότι ξέρετε τι συνέβη με τον πρώην Επίτροπο, τον κύριο Ντάλι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο, φαίνεται πως όχι. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Ερμάν Φοντιέ από πλευράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων. Μαγκίνες, κάτι το άσχετο και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το διασαφηνίσετε τώρα, θα ψηφίσουμε το Μάρτιο για θέματα αναθεώρησης της ΚΑΠ. Ε, από όσο γνωρίζετε Πότε ακριβώς θα ξέρουμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία το Μάρτιο. Το θέμα θα το δούμε αύριο όταν μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν θα γίνει τελική ψηφοφορία, από όσο γνωρίζω, για τα τέσσερα μεγάλα νομοθετήματα, η τελική ψηφοφορία θα σχετίζεται με, την, με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή, τότε θα ψηφίσουμε το Μάρτιο μόνο την εντολή διαπραγμάτευσης που επιβεβαιώνει όχι μόνο τη δική μας ψηφοφορία, του συμβιβασμούς αλλά και όλες τις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι ομάδες με καταβούληση ψηφοφορία. Στη συνέχεια θα δούμε πώς διαγράφεται η μελλοντική μας στρατηγική με βάση τις ε, πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές διότι και την προηγούμενη Δευτέρα στη συνάντηση Σούλς Βαν Ρομπόι και Μπαρόζο υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία και εκφράστηκαν και επικρίσεις ως προς τη συμφωνία αυτή. Θα δούμε λοιπόν πώς διαγράφεται το μέλλον, ποιες θα είναι οι αποφάσεις και θα υπάρξει και μια πρόταση ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε κατά την Ολομέλεια του Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπω γιατί πρέπει να αλλάξει η μερίσια διάταξή μας και η ατζέντα μας γενικότερα, διότι μιλάμε για μια εντολή διαπραγματεύσεων που θα ψηφιστεί κατά την επόμενη Ολομέλεια. Δίνω το λόγο στον Χέρμαν Φοντιέ από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας Τροφίμων που θα μας μιλήσει για αυτή τη μελέτη και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις ε, παρεμβάσεις των μέλων. Έχετε το λόγο. Herman Fontier, pronto? Qualche problema tecnico? Yeah, there's a small problem. I don't see the presentation. Ah, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, δεν βλέπω την παρουσίασή μου στην οθόνη μου. Είναι ένα προβληματάκι αυτό. Okay. Um, good afternoon. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε στη συνεδρίαση αυτή ε, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της ΕΦΣΚΑ για τη μελέτη σχετικά με τα νεονικοτινοειδή εντομοκτών. Πήραμε εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να σας ε, τονίσω ορισμένα στοιχεία κλειδιά. Ε, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη μέχρι ε, τέλη του προηγουμένου έτους, όπως και πράξαμε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ε, ποιες ήταν οι ουσίες που έπρεπε να εξετάσουμε. Η μηδακλοπρίδη, κλωθιανιδίνη και θιαμεδοξάμι που εγκρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα τρία άλλες δύο μάλλον ουσίες που είναι λιγότερο τοξικές για τις μέλισσες δεν μας έχουν αναθέσει εντολή να τις εξετάσουμε. Για τα τρία νέα νοικοτινοειδή λοιπόν που μας ανάθεσαν, μας, είδα, μας ζήτησαν να κοιτάξουμε ε, τι γίνεται με τη χρήση του σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης μας υπέδειξε ποια στοιχεία έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Ε, εκείνοι που ζητούσαν την έγκριση της δραστικής ουσίας και τα κράτη-μέλη για να δοθεί η άδεια κυκλοφορίας των δραστικών αυτών ουσιών. Μας ζήτησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε ένα κείμενο ε, το οποίο είχε προετοιμάσει το αντίστοιχο πάνελ της ΕΦΣΑ για τα ε, προϊόντα φυτοπροστασίας και πώς δρούν στις μέλισσες. Αυτή η επιστημονική γνωμοδότηση είναι το πρώτο βήμα προς ε, την εκπόνηση και τελικά έγκριση ενός κειμένου κατευθυντηρίου γραμμών της ΕΦΣΑ για να δούμε ποια θα είναι η μεθοδολογία για τις μέλισσες. Αυτό το κείμενο ε, πρόκειται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2013 από την ΕΦΣΑ. Είπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΦΣΑ, να λάβετε υπόψη σας και όλες τις άλλες ε, σχετικές μελέτες ε, που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση, την έρευνα. Τι κάναμε λοιπόν, ποια ήταν η μεθοδολογία μας για να καταλήξουμε. Ε, στην αρχή συλλέξαμε στοιχεία και από τα κράτη-μέλη και από εκείνους που ζητούσαν έγκριση των προϊόντων για να συγκεντρώσουμε όλες τις μελέτες. Συλλέξαμε όλη την πληροφορία που υπάρχει καταρχώς από τα κράτη-μέλη ε, τη βιβλιογραφία που έχει δημοσιευθεί, καθώς επίσης και ε, τα στοιχεία παρακολούθησης και ελέγχου τα κράτη-μέλη. Ε, καλέσαμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να μας δώσουν ό,τι στοιχεία είχαν και από τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνωμοδότηση του πάνελ μας, σωματώσαμε όλα τα νέα επιστημονικά στοιχεία, γιατί αυτή η επιστημονική γνωμοδότηση εμπερίχε κάθε νέα δημοσίευση στη βιβλιογραφία ως ένα πρώτο σχόλιο. Το πάνελ αυτό που ονομάζεται PPR ε, έχει λάβει υπόψη του την πρόσφατα δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία για τις επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στις μέλισσες. Λοιπόν, λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση κινδύνου και τα νέα επιστημονικά στοιχεία, ας πούμε για τα μελίσια και πώς αυτά αναπτύσσονται ε, και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Όλα αυτά ε, έχουν ενσωματωθεί στην επιστημονική γνώμη. Έχουμε αξιολογήσει όλα τα στοιχεία λοιπόν που ε, συλλέξαμε και με εκτίμηση κινδύνου και για τον οξύ κίνδυνο και για το χρόνιο κίνδυνο και διάφορες επιπτώσεις που δεν οδηγούν στο θάνατο πάντα των μελισσών. Ε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της σποράς, ε, οι ε, σπόροι αυτοί ενδεχομένως να εκπέμουν κάποια σκόνη ή μικροσωματίδια. αυτά τα εξετάσαμε την έκθεση των μελισσών και επίσης τα κατάλοιπα σε νέκταρ και σε γύρι των καλλιεργειών που έχουν ψεκαστεί με αυτά τα εντομοκτώνα. Και επίσης ε, ε, μετρήσαμε και τι ε, γίνεται στα ζυζάνια. Και η τρίτη μελέτη αφορούσε και στην εφίδρωση μελετήσαμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό. η, τα φυτά στα φύλλα τους βγάζουν σταγόνες νερού και πολύ μικρές σταγόνες που μπορεί να περιέχουν ε, πολύ μεγάλη συγκέντρωση νοικοτινοειδών. Ε, Έχουμε λοιπόν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Συνημένα με τα συμπεράσματα υπάρχουν και κάποιες σημειώσεις για την αξιολόγηση της μελέτης. Για κάθε ε, μελέτη που αξιολογήθηκε. Δηλαδή είναι τελείως ε, διαφανής ε, και διαυγής αυτή η διαδικασία και τα συμπεράσματα είναι στη διάθεσή σας. Εάν θέλετε να κατανοήσετε πλήρως ε, τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε στις μελέτες αυτές και τη μεθοδολογία μας. Το σχέδιο συμπερασμάτων έχει διαβαστεί ε, στις αρχές αρχές των κρατών μελών και τους ζητήσαμε να μας κάνουν κάποια σχόλια ε, για ε, τα συμπεράσματα αυτά. Βάσει ε, των σχολείων που λάβαμε στη συνέχεια έγινε μια συζήτηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων, εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη που έχουν ορίσει οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Then after that meeting... Μετά τη συνεδρίαση αυτή, τελικά καταλήξαμε σε συμπεράσματα που είναι ανεξάρτητα, καθότι είμαστε ανεξάρτητος επιστημονικός ε, οργανισμός. Στις 19 Δεκεμβρίου υιοθετήθηκαν αυτά τα συμπεράσματα. Με λίγα λόγια, πού καταλήξαμε δεν είχαμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την εκτίμηση κινδύνου. Θα επανέλθω σε αυτό στο τελευταίο. Ε, ε Έχουμε αναφέρει στα συμπεράσματά μας όλα τα κενά στα δεδομένα ε, και όλες τις αβεβαιότητες που συνδέονται με την εκτίμηση κινδύνου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για λόγους διαφάνειας. Δεν είχαμε επαρκή στοιχεία για να καταλήξουμε και οι διαχειριστές και αναλυτές κινδύνου θα πρέπει να κατανοούν πλήρως ε, τα επίπεδα ανασφάλειας που μας διακατέχουν λάβαμε υπόψη όλες τις χρήσεις και για κάθε χρήση ε, δώσαμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μας σε πολλά ε, στοιχεία. Και τι μπορεί να είναι αυτό. Ότι μπορεί να είχαμε μεν αρκετά στοιχεία για την ε, ανάλυση κινδύνου και τελικά καταλήξαμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει να σας πω ότι καμιά φορά ο κίνδυνος που εντοπίστηκε είχε να κάνει με ένα πρώτο στάδιο ανάλυσης κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό. Σε περίπτωση που υπήρχε υψηλότερος κίνδυνος ή άλλη μελέτη πιο πλήρης ή ε, κατάληξη και το συμπέρασμα μπορεί να ήταν διαφορετικό ως προς την ανάλυση κινδύνου. Δεν είχαμε όμως υψηλότερου επίπεδου μελέτες και χρησιμοποίησαμε ε, το, πρώτο βαθμό, ας πούμε, first tier λέγεται αυτό στα αγγλικά, ε, εκτίμησης κινδύνου. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε, γιατί είτε δεν είχαμε αρκετά στοιχεία, είτε δεν είχαμε ε, τον τρόπο να εκτιμήσουμε σωστά τον κίνδυνο. Ε, ε, οπότε ε, αναφέρουμε ότι υπάρχουν κενά και προβλήματα. Και τέλος υπήρξε και κατάσταση όπου για ορισμένες εκτιμήσεις κινδύνου μπορέσαμε να καταλήξουμε και καταλήξαμε σε αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν υπήρχε κίνδυνος. Ας πούμε, σε ζαχαρότευτλα η έκθεση των τεύτλων. Συμπέρασμα λοιπόν και συνοψίζω με δύο λόγια η έκθεση σε γύρι και νέκτα Χαμηλού κινδύνου ήταν τα φυτά που δεν ήταν ελκυστικά για μέλισσες αλλά για άλλες χρήσεις τι σημαίνει αυτό. Είτε έχει εντοπιστεί κίνδυνος είτε ε, ήταν ανεπαρκή τα στοιχεία για να καταλήξουμε και να ολοκληρώσουμε την ανάλυση κινδύνου. Η έκθεση στη σκόνη. Ε, κίνδυνος για τις μέλισσες υπήρχε ή δεν μπορούσε να αποκλειστεί με κάποιε κάποιες εξαιρέσεις ε, όπως αφορά τα ζαχαρότεφλα ή τις καλλιέργειες ε, σε θερμοκήπια ε, ή τη χρήση ορισμένων ειδικών σπόρων. Η έκθεση στην εφίδρωση αφορούσε μόνο αραβόσιτο που είχε υποστεί επεξεργασία με θεία μεθοξάμι και αυτό είχε πραγματικά οξία επίπτωση στις μέλισσες. Συνοψίζω. Ποιο είναι ο κίνδυνο, λοιπόν, για τους οξείς κίνδυνους, όχι τους χρόνιους. Ε, εφίδρωση, γύρι και νέκταρ για τις τρεις ενεργές δραστικές ουσίες. Συγγνώμη. Έτσι αξιολογήσαμε, ολοκληρώσαμε τη μελέτη και εντοπίσαμε τον κίνδυνο. Ε, για την χλωθιανίδη ε, η σκόνη έχει να κάνει με τα δημητριακά, τον αραβόσιτο και κάποιους άλλες καλλιέργειες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια είχαμε ε, ένα κίνδυνο μακροπρόθεσμο που δεν μπορούσαμε να το μελετήσουμε γιατί δεν είχαμε αρκετά στοιχεία για μακροχρόνια εξέλιξη των ε, ε, μελισσιών και δεν ξέραμε ποιος είναι ο κίνδυνος για άλλα έντομα που κάνουν την επικονίαση και δεν είναι μέλισσες ανάλογα με την καλλιέργεια η καλλιέργεια εκτός από ότι τα εντομοκτώνα μπορεί να έχει επιμολυνθεί με άλλα στοιχεία από το έδαφος. Ε, Επίσης υπάρχει ε, κίνδυνος ε, και από άλλα ε, εντομοκτώνα από άλλες ουσίες, αλλά επαναλαμβάνω δεν είχαμε πάντα ε, όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας για να αποκλείσουμε ή να ε, καταλήξουμε σε κίνδυνο. Επίσης υπάρχει κίνδυνος από την έκθεση σε δόσεις που δεν προκαλούν το θάνατο, υπάρχει κίνδυνος από την εφίδρωση των φυτών και γενικότερα αν δεν απατώμε από τον αραβόσιτο όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισήγηση. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω εξ ονόματος της Επιτροπής μας τον ε, Περιφερειακό Υπουργό, τον κύριο Κάμπριελ Κόμπαν, τον ε, Βαλερή των Νήσων και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε μαζί μας κύριε Υπουργέ είδα ότι είναι, διαπίστωσα είναι πολύ εγγεγραμμένη επειδή είναι τεχνική η η εισήγηση αυτή της ΕΑΤ. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα μιλήσουν ως προς θέματα πολιτικής υφής και εμβέλειας και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας και τον Επίτροπο Βότς. Θα ήθελα να είσαστε συνοπτικοί, διότι υπάρχουν 15 εγγεγραμμένοι ομιλητές. Ο κύριος Στέρντι καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στην Επιτροπή αυτή. Ε, με ανησυχεί πολύ ο τρόπος που έγινε η παρουσίαση αυτή. Διότι ο μιλητή έλεγε συνέχεια ότι δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε, υπάρχουν κενά στι πληροφορίε, το έλεγε συνέχεια. Είναι λοιπόν σοβαρό το θέμα αυτό και όπω και ο κύριο Σεμποβέ θα πρέπει να εξηγήσω γιατί βρίσκομαι εδώ. Είμαι ε, Πρόεδρο ε, τη Ένωση Μελισσοκόμων του Κέμπριτ και τυχαίνει να είμαι και αγρότη. Οπότε ε, με ενδιαφέρει για δύο λόγου το θέμα αυτό με ανησυχεί η ταχύτητα εφαρμογής ε, της ε, πρότασης αυτής. Ε, Ιούνιο 2013 αναφέρονται πρότυπα τα οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα. Μου φαίνεται ότι όλοι βλέπουμε όλη την κατάσταση χωρίς να δούμε το πλαίσιο. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι να απαγορεύσουμε ένα προϊόν για τα οποία δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να πρέπει οι γεωργοί να πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλο προϊόν το οποίο ε, να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις ε, μέλισσες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να σταματήσουμε εδώ και να έχουμε μια σωστή μελέτη των επιπτώσεων. Κέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχετε δίκιο. Μιλάτε στους λάθος ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Εγώ τις περισσότερες ερωτήσεις που θέλω να θέσω θέλω να τις, ερωτήσω, θέλω να τις θέσω στην Κομισιόν, διότι ε, οι δράσεις της Κομισιόν είναι το πρόβλημα εδώ, αλλά ε, κάποιες παρατηρήσεις προς την ΕΦΣΑ. Ε, Είπατε ότι ασχολείστε με ε, τις ε, νέες κανονιστικές απαιτήσεις επάνω σε ένα ε, έγγραφο το οποίο θα εκδοθεί τον Μάιο. Μπορείτε να μας πείτε εάν, είναι, εάν ενδείκνεται η απαγόρευση δεδομένου ότι δεν έχει καν εγκριθεί το έγγραφο ακόμα. Εσείς υποθέτετε ότι θα εγκριθεί και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω γιατί η ΕΦΣΑ υποβάλει σύσταση ε, τη, τη, στιγμή που δεν υπά... για, για, το folio treatment ε, για το οποίο δεν έχουμε καθόλου ε, στοιχεία. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει ήδη μια επιστημονική ανάλυση. Η κυρία Αγιούσου και μετά Άγνιο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και την ΕΑΤ για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε και για την ειλικρίνεια που την ε, διακατέχει λέγοντας ότι δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία για μια πραγματική αξιολόγηση. Αυτό είναι και το πλέον ε, σημαντικό. πέρα από τις άλλες επιπτώσεις των νέων οικοτινοειδών εντομοκτώνων. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι, ε, με ενδιαφέρει το ζήτημα γιατί εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος ε, παραγωγέας ε, μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για μια μεγάλη εξαγωγή και γι' αυτό αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να δούμε ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε συστάσεις τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι για την επιστημονική βάση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Φήμων κατά πόσο έχουν συνεργαστεί με την Ισπανία, γιατί στην Ισπανία έχουμε ένα ε, ερευνητικό κέντρο, το Μαρία Νοηγές, το οποίο έχει ε, δημοσιεύσει μία μελέτη που ακριβώς ασχολείται με την φάση επικονίασης και τις επιπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν. Στις μελέτες αυτές, οι μελέτες αυτές ε, δείχνουν ότι ε, το γύρι που υπάρχει στις κυψέλες τα, δεν υπάρχουν ε, υπολείμματα νεονικοτινοειδών πάρα, πάρα πολύ λίγα, δηλαδή ανέρχονται σε ένα 1%. Και οι μελισσοκόμοι ανησυχούν ιδιαίτερα για την ύπαρξη αυτών των εντομοκτώνων παρά το γεγονός ότι είναι αμεληταία η ποσότης τους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε δηλαδή να απαγορεύσουμε αυτό το εντομοκτόνο παρά την ύψιστη σημασία που έχει. Θα πρέπει να ξέρουμε ε, κατά πόσο μπορεί να ισχύσει όχι αυτή την, η πρακτική και νομίζω ότι προτρέξατε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. άγνιο. μετά Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα ανακοινωθέν τύπου νομίζω θα οδηγήσει πανικό, ε, κάτι που έχω δει στη Γεωργία τουλάχιστον πέντε φορές. Ε, άκουσα κάποτε έναν πολιτικό να κάνει μια ε, αρνητική δήλωση για τη σαλμονέλα και τα αυγά που τελικά ήταν αβάσιμη. Είδαμε ένα σωρό τεστ. Κάποιοι Είπαν ότι χιλιάδες ε, θα έπρεπε να πεθάνουν λόγω ε, της σε εγκεφαλοπάθειας. Ε, ακόμα δεν έχει πεθάνει κανένας. Για τα γενετικά τροποποιημένα λέγανε εκατομμύρια άνθρωποι τρώνε τέτοιες τροφές χωρίς να έχουν πάθει ούτε πονόκυλο και οι γεωργοί ξοδεύουν ένα σωρό χρήματα προσπαθώντας να αλλάξουν το, το, το καιρό και συνέχεια ξοδεύονται χρήματα για μη υπαρκτά προβλήματα. Μπορεί ε, τα νεονικοτονοειδό να αποτελέσουν πραγματικό πρόβλημα, αλλά για να πιστώ θα ήθελα να δω πρώτα ε, αποτελέσματα από μια δοκιμή σε ε, ε εκμετάλλευση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ξέρω ότι ε, θα γίνει αντικειμενικά. Ε, νομίζω πολύ συχνά μας συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και δεν χρειάζεται. Κύριε κυρία Ντελάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς η μελισσοκομεία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της γεωργίας και μπορούμε να συζητάμε χρόνια ολόκληρα για επιστημονικά δεδομένα και να βρούμε και ένα λόγο ε, που δεν είναι 100% κάτι σίγουρο, αλλά μόνο 99%. Τούτων λεχθέντων όμως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία όπως ε, ε, παρουσιάζει η ΕΦΣΑ. Την ΕΦΣΑ δεν τη δημιουργήσαμε γιατί έτσι έχει δουλειά και η δουλειά της είναι να κάνει κάποια πράγματα, είναι εμπειρογνώμονες και οι πολιτικοί δεν τα γνωρίζουν αυτά και θα πρέπει να μας συμβουλεύουν οι εμπειρογνώμονες. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, όσο γίνεται πιο κοντά στη γνωμοδότηση και στι συμβουλέ τη ΕΦΣΑ. Και υπάρχουν κάποιε. Ε, περιπτώσεις ε, που δεν ισχύει αυτό. Ας πούμε, ε, η επεξεργασία των σπόρων. Σωστά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση για τις καλλιέργειες για τα φυτά που προσελκύουν τις μέλισσες. Δηλαδή είναι τα δημητριακά και ο αραβόσιτος. Κάποιος βουλευτής θα ζητήσει ε, βέβαια και άλλη μελέτη, αλλά νομίζω προσωρινά χρειάζεται απαγόρευση για αυτά τα φυτά που προσεκύουν μέλισσες. Υπάρχουν όμως και τα ζαχαρότεφλα που δεν τραβάνε τι μέλισσες. Αυτό θα πρέπει να είναι εξαίρεση. Η ε, χρήση ε, τέτοιων προϊόντων για προϊόντα φυτοπροστασίας θα πρέπει βέβαια να περιορίζεται ε, ή αν υπάρχει δυνατότητα ε, να υπάρχει επεξεργασία των σπόρων όταν δεν ε, πρόκειται για μέλισσες είναι καλύτερο γιατί δεν έρχεσαι μετά να ψεκάζει τα φύλλα και το φυτό. Αλλά όταν είναι κλειστό το περιβάλλον σε θερμοκήπια, πολύ σωστά λέει η Εύσα, δεν υπάρχει κίνδυνος ή τουλάχιστον περιορισμένος. Αλλά δεν βλέπω επιστημονικά στοιχεία να τα λαμβάνει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο ε, ας πούμε για ε, φυτά που ε, έχουν ανθοφορήσει ε, όπως είναι το κουνουπίδι ας πούμε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση που δεν είναι στο στάδιο του πράσινου φυτού και των φύλων. Λοιπόν, προστασία φυτοπροστασία με επεξεργασία σπόρων να απαγορεύεται όταν πρόκειται για φυτά που προσελκύουν τις μέλισσες. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό ούτε στα ζαχαρότευτλα ούτε στα θερμοκήπια που δεν ενέχονται οι μέλισσες. Εγώ είμαι πρόθυμη να σκεφτώ και να ακολουθήσω και τη γνωμοδότηση και τις συμβουλές που εμείς ζητάμε από την ΕΦΣΑ την οποία εμείς φτιάξαμε για μας. Η κυρία Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι τα συμπεράσματα της σημερινής μελέτης καταδεικνύουν ότι πραγματικά ε, ενυπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις ε, ε, μέλισσες από τη χρήση αυτών των νεονικοτινοειδών εντομοκτώνων. Τώρα, με βάση αυτά που ελέγχθησαν και πριν φτάσουμε σε ε, απτά συμπεράσματα, ο, ο κύριος Στέρντι αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε αμφιβολίες για την βιωσιμότητα αυτής της μελέτης και για τη σκοπιμότητα, με συγχωρείτε, για τη σκοπιμότητα αυτής της μελέτης. Λείπουν πολλά στοιχεία. Η μελέτη είναι ελλειπής και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε πραγματικά αυτή τη μελέτη. Ποιος είναι ο βαθμός ασφάλειας ή μη ασφάλειας των συμπερισμάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω την τάση να πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία μελέτη η οποία ε, οδηγεί σε μία κινδυνολογία αλλά τι κινδυνολογία. Είναι κατακαιρματισμένη και δεν έχει ε, επιστημονικά αμυγή, επιστημονικά στοιχεία. Σε σχέση τώρα με τη σημασία των μελισσών στη Γεωργία, το θέμα είναι απόλυτα σαφές, δεν το αμφισβητεί κανείς. Το 91 μιλούσαμε για ουσίες που ήταν επικίνδυνες που ανέρχονταν σε χίλιες. Τώρα είναι 250, δηλαδή έχει συρρυκνωθεί, έχει μειωθεί ο αριθμός τους. Αλλά δεν προβάλλονται και άλλες εναλλακτικές λύσεις ή επεξεργασίες των ε, σπόρων Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα εποπτείας και αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολήσει είναι και, άλλοι, και άλλες σειρές Πέρα από αυτή τη μελέτη η οποία υποβλήθηκε εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ή κάποιος άλλος φορέας θα προβάλλει μία άλλη μελέτη για τη μείωση της ε, τοξικότητας κατά την επεξεργασία ε, φυτών στη γεωργία. Γιατί σήμερα έχουμε μία ουσία, αύριο θα έχουμε μία άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι να απαλύνουμε τους ε, κινδύνους και αυτό ακριβώς θα πρέπει να απασχολεί πρωτίστως και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμου. Όσλινγκ και μετά Σμιτ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκπλήσουμε λίγο τώρα που όλοι μιλούν αρνητικά για τη μελέτη της ΕΦΣΑ και ε, φωνάζουν για τις οικονομικές απώλειες της γεωργίας. Μα έχουμε σαφές ε, μελέτες ότι αυτά τα προϊόντα είναι επιβλαβή για τις μέλισσες. Στη Γερμανία έχουν χαθεί ολόκληροι πληθυσμοί μελισσών. Δεν θα πρέπει να αποδείξουμε ε, ότι υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος. Και μια παλιά αρχή της Ένωσης είναι όταν υπάρχει αμφιβολία επιλέγουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων και την ασφάλεια ε, των ε, μελισσών που είναι από τα πιο παραγωγικά και πιο χρήσιμα στη γεωργία και στις ζώα. Τώρα διάβασα όλη τη μελέτη της χημικής βιομηχανίας που έχει παράλογα στοιχεία για την απώλεια της γεωργίας υποτιθέμενα. Αλλά από ό,τι φαίνεται ε, ε, για τη μελέτη της ΕΦΣΑ όλοι αμφιβάλλουν και βέβαια υπάρχουν κενά και ελλείμματα και τίποτα δεν έχουν ε, μελετηθεί και ερευνηθεί 100%. Από την άλλη έχουμε πάρα πολύ σαφείς ενδείξεις ότι χάσαμε 50% του αποθέματος μελισσών. Και δεν φταίει μόνο η βαρόαση και τα παράστα και αρρώστιες το μέλισσον, αλλά είναι τα εντομοκτώνα, ε, ε, είναι τα φυτοφάρμακα και άλλα φάρμακα και θα πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Τι θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόδειξη ότι υπάρχει κίνδυνος και να έχουμε 33 μελέτες που να μας το αποδεικνύουν μπορεί να έχουν χαθεί μέχρι τότε μέλισσες. Ε, θα πρέπει και με την αρχή της προφύλαξης να προχωρήσουμε και τα μέτρα ε, πέρα από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν έγινε και τίποτα αν απαγορεύσουμε τρεις ουσίες. Δεν μπορούμε στην Επιτροπή ε, της Γεωργίας να είμαστε πάντα στο πλευρό της χημικής βιομηχανίας και των χρηστών αυτών των φυτοφαρμάκων και να μην σκεφτόμαστε και τα συμφέροντα για εκείνων που ε, θεωρούν σημαντικές τις μέλισσες, γιατί είναι, είναι από τα σημαντικότερα έντομα και ζώα πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω τα στοιχεία της ΕΦΣΑ και να πω ότι χρειαζόμαστε να λάβουμε και περαιτέρω μέτρα και πιο ισχυρές απαγορεύσεις να επιβάλλουμε. Grazie Martin ε, Schmidt. Adam e Martin Schmidt, Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, θα ε, παναλάβω αυτά που είπαν άλλοι συνάδελφοι, αλλά ε, εμένα μου αρέσει η προσέγγιση Λάγκ, την βρίσκω πολύ ισορροπημένη. Ε, ε, επίσης, θα ήθελα να επενέσω τον συνάδελφο από την ΕΦΣΑ για μια ε, επιστημονικά τίμια ε, προσέγγιση και αυτή η διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και την πολιτική. θα πρέπει να προσέξουμε η επιστήμη να μην γίνεται θέμα θεολογίας τελικά, αντί για να είναι αντικειμενική εξέταση των γεγονότων. Έχω συζητήσει με επιστημονικό σύμβουλο πώς ενσωματώνουμε τα θέματα της επιστήμης στην πολιτική. Ε, και το, σήμερα ακούμε στοιχεία τα οποία δίδονται σαν να είναι οι δέκα εντολές. Ε, χωρίς να έχουμε εξετάσει από πού προέρχονται και ποιοι είναι οι στόχοι. Η ΕΦΣΑ είναι η μόνη αντικειμενική υπηρεσία από την οποία έχουμε στοιχεία σχετικά με το θέμα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ε, αποδεδειγμένο ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι ζωτική σημασία για τη γεωργία μας αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των ε, χημικών αυτών και νομίζω ότι η ε, Κομισιόν έχει ενεργήσει ρεαλιστικά και αναλογικά. Ε, το ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνε ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μα σταματήσουν να το να δράσουμε, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Εύσα τι άλλε έρευνε κάνετε πάνω σε αυτό, διότι σίγουρα δεν πρόκειται για το τέλο ε, τη συζήτηση αυτή. Είμαι υπέρ τη προσέγγιση τη Κομισιόν. Προσωπικά πιστεύω θα πρέπει να πάει ακόμα πιο πέρα, αλλά χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να μην, έρχονται, να προέρχονται από λόμπι με συγκεκριμένα ε, οικονομικά συμφέροντα. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Εύσα είναι τι υπεραιτέρω δουλειά κάνετε πάνω σε αυτό. Και θα δεχόσασταν μια σειρά ερωτημάτων από την Επιτροπή μας σχετικά με τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Γκαρθία Πέρες, συμμερίζομαι το γεγονός ότι αυτό που θα πρέπει να δούμε πρωτίστως είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα σε σχέση με τις εφαρμογές, την εφαρμογή αυτού του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο μπορούμε να δούμε και με τον Επίτροπο μεταγενέστερα σε σχέση με την εισήγηση που έγινε, για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις. Συμφωνώ ότι έχει ήδη εκφραστεί ανησυχία σε σχέση με την κατάσταση της μελισσοκομείας στην Ευρώπη, το γεγονός ότι εξαφανίζονται πολλές κυψέλες και χρειαζόμαστε επιστημονικά στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι επίσης γεγονός ότι η ΕΦΣΑ, και εδώ μιλώ αντικειμενικά, γιατί βασίζομαι στην αρχική εισήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, έθιξε λοιπόν η ΕΦΣΑ δύο ζητήματα που μας απασχολούν. Μιλήσαμε για τη χρήση της μεθοδολογίας είναι μια μεθοδολογία η οποία δεν θα ισχύει από το Μάιο και μετά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η νέα μεθοδολογία, η οποία ακόμα δεν έχει εγκριθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειραγώγηση αυτών των στοιχείων ή κακομεταχείριση. Υπάρχουν κενά, αμφιβολίες, μη διάθεση πολλών στοιχείων, έλλειψη στοιχείων. Καταλαβαίνουμε ότι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια η ΕΦΣΑ γιατί είναι ένας ανεξάρτητος και επιστημονικός οργανισμός, αλλά θα θέλαμε να μπορέσει να ανταποκριθεί επιστημονικά έτσι ώστε εμείς στη συνέχεια να μπορέσουμε να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις. Θεωρείτε ότι είχατε αρκετό χρόνο για να διενεργηθεί μία σοβαρή μελέτη, χρειάζεται και άλλη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Θα ήθελα ο κύριος Φοντιέ να μου απαντήσει στα δύο αυτά ερωτήματα. Κώστιντζερ και μετά George Lyon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ για την παρουσίαση της μελέτης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι μέλισσες αποτελούν ε, απαραίτητο κομμάτι ε, της υπαίθρου μας ε, και όταν έχουμε τόσο μαζικά στοιχεία και δεδομένα όταν βλέπουμε να πεθαίνουν έτσι οι θα πρέπει να εξάγουμε τα σωστά πολιτικά συμπεράσματα. Δεν έχω δει καμία μελέτη της χημικής βιομηχανίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί με βάση μια τόσο ελλειπούς έκθεσης θα πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερα με εκπλήσει ότι στην έκθεση της ΕΦΣΑ αναφέρονται εκθέσεις που μάλλον δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μελέτες ε, που δεν δείχνουν να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο, στο, ε, στο θάνατο των μελισσών ε, και τα νέων και το είδη. στην Αυστρία βλέπουμε να πεθαίνουν μέλισσες σε, σε περιοχές όπου δεν έχουμε ε, ε, μαζική γεωργία και χρήση νεονικοτινοειδών. Γι' αυτό... θα ήθελα να πω ότι στην Αυστρία εδώ και χρόνια έχουμε σχετικό πρόγραμμα, το Μελίσσα και... Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εκθέσεις αυτές που ανέφερα εδώ. Σίγουρα πεθαίνουν οι μέλισσες, υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε επίσης ε, στην Αυστρία επειδή είναι τόσο μικρές ε, οι καλλιέργειες να έχουμε αμεψή σπορά. Ε, κάποιοι θεωρούν ε, εναλλακτική λύση τη, τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους ε, και πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ε, στην Αυστρία ήδη έχουμε εφαρμόσει πολλά μέτρα, όπως για παράδειγμα ε, όχι χρήση των ε, διαφόρων ουσιών ε, ε, ε, κατά την, σε κάποιες εποχές του έτους, την αμυσισφορά όπως είπα. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε μέτρα θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή επιστημονική βάση. Θα ήθελα να ακούσω από τον εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ πώς η ΕΦΣΑ δημοσιεύει τόσο ελλειπή και γιατί δεν περίμενε ώστε να έχει το χρόνο να μελετήσει εις βάθος το πρόβλημα αυτό. Και θα ήθελα να αναφέρω και μία ακόμα πτυχή όσον αφορά το ότι πεθαίνουν μέλη σε περιοχές όπου δεν χρησιμοποιούνται ε, νεονικοτινοειδή. Έχουμε μελέτες ε, σχετικά με την ε, διασταύρωση ευρωπαϊκών μελισσών με αμερικάνικες. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η ΕΦΣΑ έχει συλλέξει στοιχεία σχετικά με το αν αυτό έχει οδηγήσει σε προβλήματα στις μέλισσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζος Λάιον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΦΣΑ για την παρουσίαση της Διάβασα τις πολλές πολλές σελίδες ε, της έκθεσης και όταν έφτασα στο τέλος είχα περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι απαντήσεις, ε, διότι παντού λέει ότι ε, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Αυτό ανακύπτει συνέχεια. Βέβαια είναι θεωρητικό το θέμα. Δεν έχουμε στοιχεία από κάποιο πείραμα ή από κάποια επιστημονική δοκιμή και είπαν ότι πιθανότατα να υπάρχει θεωρητικό πρόβλημα. Ε, αλλά βέβαια θα πρέπει να το πάρουμε αυτό σοβαρά. Αλλά θεωρητικός κίνδυνος ε, και πραγματική ζημιά στις μέλισσες είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν βλέπω να υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο λόγω των λοιπόν στοιχείων που αναφέρουν και την έλλειψη σχετικών μελετών. Για παράδειγμα, δεν έχουν εξεταστεί οι αρινές καλλιέργειες, ε, διότι είναι πολύ διαφορετικές από τις χειμερινές. Ε, διότι το χειμώνα παίρνει κανείς ε, σε, εποχή που οι μέλισσες βρίσκονται μέσα στα μελίσια θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την, ε, ε τις μεθόδους ε, ποτισμού των σπόρων ε, κατά το χειμώνα. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα, αλλά αναρωτιέμαι εάν η ανταπόκριση που προτείνεται δικαιολογείται με βάση τα στοιχεία που έχουμε σήμερα. αυτό βέβαια δεν είναι ερώτηση προς την ΕΦΣΑ. ερώτηση προς την ΕΦΣΑ είναι δεδομένων των κενών που υπάρχουν στα δεδομένα τι θα πρέπει ακόμα να γίνει για να μπορείτε να σε καταλήξετε σε καλύτερα συμπεράσματα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μιλάμε για πραγματικούς κινδύνους. Και δεύτερον, τι δουλειά πρέπει να γίνει σε πρακτικό επίπεδο για να αξιολογηθούν οι συνέπειες στους πληθυσμούς των μέλισσών, διότι άλλο είναι ο θεωρητικός κίνδυνος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόση ζημιά υφίστανται οι πληθυσμοί των μέλισσών. Ε, καταλαβαίνω ότι μειώνεται ο πληθυσμός ε, των μελισσών, αλλά ε, έχω εδώ μια μελέτη που ε, δείχνει σημαντικές διακυμάνσεις, ιδιαίτερα στη Φιλανδία. Αυτό πιθανότατα έχει να κάνει με τους σκληρούς χειμώνες στη Φιλανδία. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορείτε να υποστηρίξετε ότι υπάρχει ευρή αναγνώριση, ότι υπάρχει σημαντική μείωση. Νομίζω ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τα στοιχεία. Σίγουρα υπάρχουν σημαντικέ διακυμάνσει όσον αφορά του πληθυσμού των μελισσών. Θα παρακαλούσα την ΕΕΦΣΑ να απαντήσει σε αυτό, διότι αυτό μα βοηθήσει να ε, καθορίσουμε τον ε, δρόμο που θα ακολουθήσουμε. Ε, κύριε Ρέιμερ, σε ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλού κυρία Η τονίζει ότι δεν έχει αρκετά στοιχεία, ούτε αριθμητικά, ούτε γενικότερα όπως είπε ο κύριο Σμιθ, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, περισσότεροι ρυθμοί, περισσότερα και, έτσι, βαθύτερα μελετημένα στοιχεία. Η ΕΦΣΑ παρόλα αυτά λέγει ότι υπάρχει κίνδυνος για τις μέλησεις και συνιστά ε, απαγόρευση ε, των προϊόντων αυτών. Νομίζω ότι είναι ακραία αυτή η απαγόρευση, ακριβώς επειδή έχουμε τόσο λίγα στοιχεία στη διάθεσή μας. Νομίζω θα πρέπει να φροντίσουμε πρώτα να βρούμε τεχνικές λύσεις. Ας πούμε, να βελτιωθούν οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη σπορά. Ε, να έχουμε, ας πούμε, στη δική μου περιφέρεια έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την κράμβη, ιδιαίτερα όταν σπέρνονται ε, το ε, χειμώνα, γιατί υπάρχει ένα παράσιτο, ένα μικρό μυγάκι που προσβάλλει αυτά τα φυτά που έχει μάλιστα τώρα αποκτήσει και αντίσταση απέναντι στο μοναδικό φυτοφάρμακο που χρησιμοποιούμε. Και ποια είναι και η ευρωπαϊκή ε, στρατηγική ε, για τις πρωτεΐνες ε, και για τις ζωοτροφές, γιατί η κραμβή είναι το μοναδικό εναλλακτικό φυτό απέναντι στη σόγια. Λοιπόν, να μην πέσουμε από τη σκύλα στη χάρευδη για να προστατεύσουμε τον ένα κλάδο να καταστρέψουμε τον άλλο. Χρειάζεται σταδιακή προσέγγιση με καλύτερα στοιχεία επιστημονικά ε, τεκμηριωμένα γιατί πολλές φορές ε, συγκρίνουμε πεπαλαιωμένα και ξεπερασμένα στοιχεία. Ακούσαμε ότι έχουν έρθει ε, μέλισσες από άλλες χώρες, έχουν γίνει διασταυρώσεις και μάλιστα υπάρχουν και αρρώστιες που επηρεάζουν. Επίσης επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή η κατάσταση. Δεν αφορά αυτό μόνο ένα εντομοκτόνο. Αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, τότε θα έχει λυθεί η κατάσταση προπολού. Ευχαριστώ. Γλάτο Φέρντερ και μετά Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι τα εντομοκτώνα είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες. Άλλωστε αυτό αναγράφεται και στην ετικέτα του προϊόντος. Ε, ποια είναι η επιτρεπόμενη δόση για να μην βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα. Αν τηρούνται αυτοί οι κανόνες και οι προδιαγραφές, τότε περιορίζεται κατά πολύ ο κίνδυνος. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα εξαλειφθεί. Δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποια ε, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ε, κάποια φυτοφάρμακα και εντομοκτώνα. Αν απαγορεύσουμε αυτές τις ουσίες και γενικότερα αυτά τα προϊόντα, ε, υπάρχουν άλλες επιπτώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουγγαρία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μελιού. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η υγεία των μελισσών. Τα εντομοκτώνα αυτά στη χώρα μας χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και πολύ στο εμπότισμα των σπόρων. Έχουμε ένα προϊόν που κυκλοφορεί από τις Ηνωμένε Πολιτείε, πάρα πολύ επικίνδυνο ε, και ε, ε, μπορεί να αφορά και το 50% του καλαμποκιού. Και, πέρυσι χάσαμε μέλισσες στην Ουγγαρία ακριβώς λόγω αυτού του προϊόντος πρωτοφανές. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτό το προϊόν στις καλλιέργειες και ε, αφάνισε τις μέλισσες. Βέβαια δεν σε ποτέ να αποδειχθεί η ε, συσχέτιση ε, της χρήσης αυτών των φυτοφαρμάκων με ε, την εξαφάνιση των μελισσών. Ε, έγινε και ένα πείραμα στην Ουγγαρία με ηλιοτρόπια. Ε, σε μια καλλιέργεια που είχε χρησιμοποιηθεί ένα νεονικό τινοειδές, δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί ότι είχε βλαβερές συνέπειες στις μέλισσες. Ξέρουμε όμως ότι χρησιμοποιούνται πλέον αυτά τα προϊόντα γιατί υπάρχουν αυτά τα παράσιτα των φυτών και στην Ουγγαρία, αλλά ε, δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί ε, ποια συνέπεια θα είχε υπαγόρευση των φυτοφαρμάκων. Θα χρησιμοποιούν τελικά άλλα προϊόντα, άλλα χημικά και άλλα ζυζανικτόνα και εντομοκτόνα... και δεν θα ε, γίνεται υπεξεργασία στο σπόρο πριν τη σπορά, αλλά θα ψεκάζουν τα φυτά και τα φύλλα τους, πράγμα που θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα για τις μέλισσες από ό,τι αν είχε υποστεί επεξεργασία ο σπόρος. Εμείς όμως στην Ουγγαρία παράγουμε και σπόρους, πολλαπλασιαστικό υλικό για ε, καλαμπόκι ας πούμε και αν απαγορευτούν αυτά τα προϊόντα θα φύγει η παραγωγή από την Ευρώπη και θα πάει στην Ουκρανία ας πούμε ή θα αρχίσουν να παράγουν γενετικά τροποποιημένο, μεταλλαγμένο καλαμπόκι ε, πράγμα που θα φέρει προς συζήτηση άλλα θέματα για τα μεταλλαγμένα. οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν αν χρησιμοποιείται σωστά ε, το κάθε προϊόν για να μπορέσουν ε, και οι γεωργοί και οι μελισσοκόμοι να ε, κανονίσουν την πορεία τους. Τελικά νομίζω ότι από νέο νοικοτινοειδή δεν χάθηκαν μέλισσες στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ε, Μακίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Εύσα για την παρουσίασή της. Είναι χρήσιμο που έχουμε αυτή την αναλυτική τεχνική συζήτηση, αλλά βέβαια η πολιτική συζήτηση τελικά θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, σχετικά με τη δεύτερη διαφάνεια, όπου η ΕΦΣΑ λέει ότι η Κομισιόν της έδωσε την εντολή. Αναρωτιέμαι εάν ήταν πολύ σύντομη η προθεσμία για να προλάβετε να αναλύσετε όλες ε, τις διαθέσιμες μελέτες. Άκουσα επίσης την ΕΦΣΑ να λέει ότι η Κομισιόν ανέφερε ποια δεδομένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η ΕΦΣΑ πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλα δεδομένα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ε, για να καταλήξει σε συμπεράσματα. Αυτό που ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι σχετικά με τα κενά στα δεδομένα ε, ε, είναι πραγματικό και θα συμφωνούσα ε, σχετικά, ε, θα συμφωνούσα στην ερώτηση η ΕΦΣΑ ε, τι προτείνει και μήπως υπάρχουν άλλα δεδομένα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θεωρητικές αναλύσεις που γίνονται στο γραφείο και τις δοκιμές που γίνονται επί τόπου. Αυτό αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους. Νομίζω ότι όλοι εδώ θέλουν να κάνουν το σωστό ώστε να είμαστε ασφαλείς. Πάντα λέγαμε ότι είναι θέμα με πολλούς παράγοντες και γι' αυτό έχω συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν η πρόταση της Κομισιόν ε, γίνει κανόνας και απαγορέψουμε... Ε, τα νεονικοτινοειδή ε, θα δούμε αύξηση στο πληθυσμό και αν ναι πότε, διότι από ό,τι κατάλαβα ε, η βαρόση είναι πολύ πιο πραγματική απειλή στην υγεία των μελισσών και ακόμα δεν έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα ε, με καθοριστικό τρόπο στην Ευρώπη. Επίσης, ε, όπως ανέφερε και ο κύριος Γκλάτφελτερ, ε, υπάρχουν ε, κάποιες συνέπειες, όπως είπε, στο δικό του κράτος μέλος. Εάν οι γεωργοί συνεχίσουν να καλλιεργούν τα προϊόντα όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα, ε, εάν έχουν καλλιέργειες όπου χρησιμοποιούνται ε, ε, αυτά τα προϊόντα, τι θα χρησιμοποιήσουν και αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανένα προϊόν, τότε ποιε θα είναι οι συνέπειε για τη γεωργία στι περιοχέ αυτέ. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, θα ευχόμουν το πρόβλημα να είναι τα νεονικοτινοειδή, διότι έτσι θα το λύναμε το πρόβλημα. Αλλά όπω ακούσαμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε κατά την επιλογή της λύσης. Διότι μπορεί τελικά η λύση να μην ταιριάζει στο πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση και ελπίζω η Εύσα να μπορεί να απαντήσει σε κάποιε από που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να πω ότι ακούσαμε πώς έχει η κατάσταση, αλλά να αρχίσουμε κάποια στιγμή να μελετούμε και τα αίτια ε, της εξαφάνισης των μελισσών. Σήμερα είδαμε μια παρουσίαση που λέγει ότι αν περιοριστούν οι ουσίες που κυκλοφορούν ή αν απαγορευτούν οι ουσίες που κυκλοφορούν, θα έχουν κάποια ε, αποτελέσματα και κάποιες επιπτώσεις. Ε, μήπως προτρέχουμε όμως. Έχουμε μελετήσει αρκετά και τα χρονικά διαστήματα που χρειάζονται. Αυτό είναι το ένα που θα ρωτήσω. Το δεύτερο. Και ποιες ουσίες θα χρησιμοποιήσουμε ως υποκατάστατα, ποιες χημικές ουσίες, σε ποιο βαθμό και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές από εκεί και πέρα στον πληθυσμό των μελισσών. γιατί υπάρχουν και ασθένειε των φυτών που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με κάποιο τρόπο, με κάποια χημικά γίνεται αυτό. Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα που είδαμε ότι καλύπτει η μελέτη. Δηλαδή, να μελετήσουμε καλύτερα και τις χώρες, τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις κλιματικές τις περιφέρειες ακόμα περισσότερο όπου επικρατούν άλλες ε, καταστάσεις σε σχέση με άλλες ε, περιφέρειες και άλλα κράτη. Δεν ξέρω πώς χρειάζεται περισσότερη εργασία εκεί από αυτού του θέματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα με προσοχή και άκουσα τα δεδομένα της μελέτης ως προς τους περιορισμούς και ως προς το βάσιμο των στοιχείων. Όλοι γνωρίζουμε τον ε, ουσιώδη ε, ρόλο των ε, επικονιαστών και το ρόλο που παίζουν στη δημόσια υγεία. Επίσης γνωρίζουμε και το ποσοστό θνησιμότητας πολλών χιλιάδων κυψελών εδώ και 20 χρόνια μετά από χρήση εντομοκτώνων. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα σε επίπεδο κοινοβουλίου και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να δούμε την επίπτωση ορισμένων προϊόντων εντομοκτώνων πριν ε, τα βάλουμε στην αγορά. Μέσα στα πλαίσια της αρχής της ε, πρόληψης θα ήθελα να αποσυρθεί αυτό το προϊόν από την αγορά όπως ε, έγινε στη Γαλλία. Να ανασταλεί τουλάχιστον η χρήση. Κάτι το οποίο στη Γαλλία ε, δεν είχε και πολύ αρνητικές συνέπειες στη Γεωργία. Αν λάβουμε υπόψη τους ενεχόμενους κινδύνους. Αν λάβουμε υπόψη αυτό τον ε, ε κίνδυνο που ελοχεύει, θα ήταν πολύ καλύτερα να προωθήσουμε μία εξειδικευμένη εργασία όπως κάνει η ΕΦΣΑ σε σχέση με το ρόλο των εντομοκτώνων και να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες έγκρισης των ε, φυτοφαρμάκων. Ευχαριστώ κύριε Στές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύντομα. Με σόκαρε λίγο αυτό που άκουσα ότι δεν μπορεί λέει να αποκλειστεί. Ωραία. Τι θα πει αυτό. Τότε να απαγορεύεται και ο χαλκός στις βιολογικές πατάτες στην καλλιέργεια γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι έχει κάποια επίπτωση στο περιβάλλον. Κάθε μέρα τρώω μέλι και θέλω πάρα πολύ να είναι τα τρόφιμά μας υγιεινά. Αλλά αυτά που ακούσαμε σήμερα για τη χρήση νέων νοικοτινοειδών με προβλημάτισαν. Τα είπε και η κυρία Έιμερς. Έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια ελαιοκράμβης στη Γερμανία και από τη δεκαετία του 60 ήμουν από τους πρώτους που έσπηρα κράμβη. Και είναι σημαντικό αυτό και μιλάμε για αμυψισπορά. Είναι πολύ σημαντική καλλιέργεια. Τι θα γίνει, δεν θα μπορούμε πλέον στην Ευρώπη να καλλιεργούμε λεοκράμβη. Θα είχαν μεγάλα προβλήματα πολλέ καλλιέργειες. Και στην αμυψισπορά είναι πάρα πολύ καλό φυτό που βελτιώνει και τη γονιμότητα του εδάφους. Και πραγματικά θα ήταν πρόβλημα εάν δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα πολλαπλασιαστικού υλικού. Και ρωτάω την Εύσα. Στη Γερμανία έχει αποδειχθεί έστω και μία περίπτωση ότι ε, ε, η επεξεργασία των σπόρων της ελαιοκράμβης προκαλεί προβλήματα σε πληθυσμούς μελισσών. Εάν ναι, να δημοσιευθεί αυτό. Βέβαια, μιλώ πάντα με τη σωστή χρήση του ε, πολλαπλασιαστικού υλικού. Υπήρξαν ίσως κάποια προβλήματα στη Γερμανία αλλά λόγω κακής χρήσης και κακών σπόρων και μη σύνομης ε, πρακτικής και συμπεριφοράς. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, είπαμε, εναλλαγή των καλλιεργειών με την άμυψη σπορά και ακριβώς επειδή από τη δεκαετία του 60 καλλιεργώ το σημεριμένο φυτό, ε, στη δεκαετία του 70 ε, είχα την ευκαιρία να καλλιεργήσω ε, μια νέα ποικιλία όταν έφτασε στη Βαβαρία και τότε εκείνο το χειμώνα που μπήκε αυτή η νέα ποικιλία ε, πάρα πολλά ζαρκάδια στη Βαβαρία. Τυχαίο ήταν αυτό. Ε, και είχε γίνει χαμός τότε στη Γερμανία ότι βγάλετε αυτό το φυτό και πέθαναν τα ζαρκάδια. Ε, όχι, κυκλοφόρησε μια ασθένεια τότε ε, μεταξύ αυτών των πληθυσμών και δεν είχε καμία σχέση με τις καλλιέργειες ε, και έχει γίνει τρομερή φασαρία ε, ότι φταίει η ελαιοκράβη. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά επιστημονικά στοιχεία και αποδείξεις αν θέλουμε να απαγορεύουμε προϊόντα και δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε κάτι όταν δεν μπορούμε 100% να αποκλείσουμε ένα κίνδυνο. Μα δεν υπάρχει αυτό. Να φύγουμε και από την αίθουσα εδώ γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι την επόμενη ε, ώρα ή τις επόμενες ώρες θα μας έρθει κανένας αστεροειδή στο κεφάλι. Ε, και μετά η Μαρία Γκάμπριελ. Θα κάνω όπως και ο κύριος Σμιθ. Κύριο Σμιθ, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός. Πρέπει λοιπόν να το πούμε γιατί είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μία αιτία για τη θνησιμότητα των μελισσών. Είναι οι ασθένειες καταρχήν, τα εντομοκτώνα και οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μία πρόσμιξη. Υπάρχουν πολλαπλές αιτίες και με τα νεονικοτινοειδή λέμε ότι πρόκειται για νευροτοξικές ουσίες οι οποίες κάνουν πλήττουν το νευρικό σύστημα των, ε, των εντόμων, των μελισσών που δεν μπορούν πια να βρουν την κυψέλη στην οποία ανήκουν και πεθαίνουν. Δηλαδή πρόκειται για ένα προϊόν που πλήττει τις μελέτες, τις, με, με συγχωρείτε, τις μέλισσες, αλλά και όλα τα έντομα επικονιαστές. Εκεί βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματος. Δεύτερον, σήμερα θεωρούμε ότι το κέρδος που δίνει στη γεωργία οι επικονιαστές είναι της τάξης των 15 δισευρώ ετησίως. Η διαδικασία επικονίασης δηλαδή. Εάν εξαφανιστούν αύριο οι μέλισσες θα υπάρχει, ε, θα υπάρχει όλεθρος, επέρχεται ένας όλεθρος και για τη διατροφή. Και τρίτο σημείο, και θα σταματήσω εδώ, στην Ιταλία, στο βορρά της Ιταλίας, υπάρχει το σχέδιο APENET, το οποίο προωθείται μέσω ε, ποράς σε σχέση με τη χρήση αυτών των εντομοκτώνων. Πρόκειται για μια επιστημονική εργασία, όπου είδαμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ζημίες, αλλά θα μπορούσαν οι παραγωγοί να μην χρησιμοποιήσουν αυτά τα εντομοκτώνα μέσα στα πλαίσια της αμυψισποράς που εισήχθη. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εύσα για την εργασία της και γιατί μας έφερε νέα στοιχεία. Πολύ συχνά άκουσα ότι δεν πρέπει να επικρίνουμε την Εύσα διότι πάντα γνωματεύει θετικά για ορισμένα προϊόντα. Για μία φορά που η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων δεν το κάνει, λέμε ότι δεν εργάζεται σοβαρά. Αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή όσοι ήταν οι υπερασπιστές της ΕΦΣΑ ε, σήμερα την κατακρίνουν. Η ΕΦΣΑ επιτέλεσε μεγάλο έργο για να είναι αντικειμενική και χαιρετίζω την εργασία της και την τιμώ. Μαρία Γκάμπριελ. Και τέλος η κυρία Λούλιν για να κλείσει αυτό το γύρο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ε, χαιρετήσω την ΕΦΣΑ για την ε, θετική εργασία ε, ως προς τα υπέρ και τα κατά αυτής της μελέτης. Όλοι ξέρουμε την ολέθρια επίπτωση των εντομοκτώνων στις μέλισσες. Αυτό είναι ευρέως γνωστό. Και σε μία μελέτη που διενεργήθηκε στη Βουλγαρία το 2011, είδαμε ότι χάθηκαν πολλές ε, μέλισσες εξαιτίας της χρήσης των εντομοκτώνων. Ένα 64% του πληθυσμού χάθηκε γιατί ακριβώς δεν υπήρχε σωστή και ρυθμισμένη χρήση των εντομοκτώνων. Οι αιτίε ε, όμως της ε, θνησιμότητας των μελισσών είναι πολλαπλές. Υπάρχει και θέμα ασθενειών, όπως είπε ο κύριος Μποβέ. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο σοβαρά το ζήτημα. Δεν θα πρέπει παρά να υπερασπιστούμε τους μελισσοκόμους και ελπίζω αυτή η συζήτηση να είναι μια συζήτηση ουσίας και να μην πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ μελιού και αραβοσίτου ή μελιού και κράμπης. Νομίζω ότι θα βγαίναμε χαμένοι όλοι από αυτή τη διαδικασία. Θα θέλαμε αυτά αποτελέσματα. Ήδη έχουν επιβληθεί περιορισμοί σε ορισμένα κράτη-μέλη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται στη Σλοβενία, την Ιταλία και τη Γαλλία που ήδη έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις, μερικώς τουλάχιστον. Θα θέλαμε να δούμε κατά πόσο μετά από αυτές τις απαγορεύσεις υπάρχουν θετικές επιπτώσεις. Επιβλήθηκε μία προθεσμία ε, δύο ετών και ξέρουμε ότι τα νεονικοτινοειδή αποτελούν έναν ενδυνάμει κίνδυνο για τα, και για τα φυτά. Γιατί μετά από δύο χρόνια μόνο γίνεται μια ανάλυση επιπτώσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εύσα για το θάρρος ε, που έδειξε θίγοντας ένα τέτοιο επώδυνο ζήτημα και να πω ότι χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα και θα πρέπει να τηρήσουμε τις προδιαγραφές ως προς τα εντομοκτώνα. Η κυρία Λούλη, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 1994 ήμουνα μόνιμη εισηγήτρια για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής μελισσοκομείας και τότε θεωρήθηκα περίγελος όταν έκανα την πρώτη εισήγηση ε, και έκθεση διότι ζήτησα βοήθεια για τη βελτίωση της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Μελισσοκομείας. Ζήτησα και μία πρημοδότηση για την ε, επικονίαση και η Επιτροπή αγνόησε αυτό το αίτημα υπήρξε ένας κανονισμός για τη βελτίωση της ε, παραγωγής και εμπορίας του μελιού. Αρχίσαμε με 10 εκατομμύρια, εκατομμύρια όχι δις και φτάσαμε σε 34 εκατομμύρια και κάθε χρόνο με είχατε υποστηρίξει και ήταν και η μόνη, η πίστοση η οποία είχε ε, αυξητική τάση παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόμασταν σε διαδικασία συναπόφασης. Χαίρομαι λοιπόν τώρα εκ των υστέρων διότι επιτέλους πολλοί συνάδελφοι ανακάλυψαν την πραγματική σημασία του ζητήματος μετά από την αυξανόμενη πνησιμότητα των ε, μελισσών. Στο ψήφισμα μας για την ε, τελευταία έκθεση για, ως προς την ε, μελισσοκομεία, συντάκτης της οποίας ήσασταν εσείς πρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν ξεχάσαμε την σημασία της μέλισσας των μελισσών στην Ευρώπη μέσα στα πλαίσια της επικονίασης. Τώρα, όταν μιλάμε για βραχυπρόθεσμη απαγόρευση ορισμένων σπόρων ή της όλης διαδικασίας χρήση εντομοκτώνων, τότε ε, αυτό θα έπρεπε να το δούμε μέσα στα πλαίσια μιας εναλλακτικής. Αν δεν υπάρχει όμως εναλλακτική, δεν ξέρω κατά πόσο, θα χάσουμε χωρίς να έχουμε αδιάσυστα επιστημονικά στοιχεία και θα χάσουν οι γεωργοί τη συγκομιδή τους. Με βάση μια γερμανική μελέτη, με βάση τα δεδομένα της Ένωσης Γεωργών, της Γερμανίας ε, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Αυτά, αυτό είχε αναφερθεί στην ε, ε, Γερμανία και δεν ξέρω κατά πόσο η ΕΦΣΑ τώρα έχει βελτιώσει ή τελειοποίησει τις αναλύσεις αυτές. Κατά πόσο υπάρχει δηλαδή μια αδιάσυστη επιστημονική βάση θα ήθελα να προσέξει η Επιτροπή. Δεν πρέπει να σπεύσει να αποφασίσει σε σχέση με την μείωση απαγόρευση ε, χρήσης σπόρων χωρίς ε, εναλλακτική. Αυτή η απαγόρευση θα οδηγούσε σε ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο η Επιτροπή θα μπορούσε να μην λάβει εσπευσμένες αποφάσεις σε επίπεδο μείωσης γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα, δηλαδή η χρήση ή μη χρήση των εντομοκτώνων. Τη στιγμή που δεν έχουμε αδειάσει στα στοιχεία ότι τα εντομοκτώνα αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικέ, αν υπάρχουν εναλλακτικές, ας τις προωθήσουμε. Αν όμως δεν υπάρχουν, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που έκανε και η Γαλλία, δηλαδή για πολιτικούς λόγους θα απαγορεύσουμε γιατί αυτό είναι δημοφιλές, ένα δημοφιλές μέτρο. Δεν θα ήταν σκοπιμότερο να βασιστούμε σε επιστημονικές αναλύσεις έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή συγκομιδή στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για άλλη μια φορά στον κύριο Έρμαν Φοντιέρ από πλευράς της ΕΦΣΑ για να μας απαντήσει στο μέτρο του δυνατού στις, ε, στα ερωτήματα που εθίγησαν και θα ήθελα να αρκεστεί στα 10 λεπτά το πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα με τον Επίτροπο Μπόρσο ο οποίος θα προσέλθει σε λίγο. Ο Χέρμαν Φοντιέρ έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεγάλη πρόκληση. Πολλές ερωτήσεις, 10 λεπτά μόνο. Ελπίζω μάλιστα να σημείωσα όλες τις ερωτήσεις που απευθύνατε προς την ΕΦΣΑ. Είχαμε μια ερώτηση σχετικά με έγγραφο καθοδήγηση, ε, γιατί ε, χρησιμοποίησαμε επιστημονική ε, γνώμη για το έγγραφο αυτό. Η απάντηση είναι απλή, η Κομισιόν μα το ζήτησε, αλλά η απάντηση είναι και κάτι παραπάνω. Γιατί η Κομισιόν μας ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε την Επιστημονική Συμβουλή, διότι η Επιστημονική Συμβουλή έχει ενσωματώσει νέα επιστημονικά δεδομένα και προφανώ η Κομισιόν θεώρησε ότι θα τα λάβουμε υπόψη μας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ότι θα λάβουμε υπόψη μας ε, την ε, νέα επιστημονική ε, φιλολογία που δείχνει τα μη θανατηφόρα αποτελέσματα στις μέλισσες. Είχαμε μία ερώτηση σχετικά με τις συστάσεις για, για τα φύλλα. Το θέμα είναι ποιος πιστεύουμε ότι είναι ο κίνδυνος. Ε, ε, δεν έχουμε υποβάλει σύσταση για την επεξεργασία των φύλων, ε, διότι δεν έχουμε εξετάσει το θέμα αυτό. Επανειλημμένα άκουσα ότι δεν λάβαμε υπόψη μας μελέτες τρίτων. Λάβαμε υπόψη μας μελέτες τρίτων σε περίπτωση όπου υπήρχαν και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, τέσσερις ε, μελέτες επιτόπου ε, έχουν δείξει την έκθεση των μελισσών στα υγρά από την εφίδρωση και αν εξετάσουμε την εθνισμότητα φαίνεται ότι η ΕΧΜΗ πραγματοποιήθηκε την στιγμή της εμφάνισης εάν Έχουμε λοιπόν μελέτες ε, πραγματικές, ε, πειραματικές, ε, θα ήθελαμε περισσότερες εάν είχαμε, αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο μελέτες που έγιναν στο γραφείο, θεωρητικές μελέτες δηλαδή. και μελέτες εργαστηρίου και ο κύριος ε, Ποβέ ανέφερε το αν έχουμε βρει τον, ε, ε, τον μόνο λόγο εθνισίμωτας των, των, των μελισσών. Ούτε λέμε ότι τα νεονικοτινοειδή είναι ο μόνος λόγος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Πιθανότατα να μπορούμε να πούμε ότι δεν αποκλείεται ότι τα νεονικοτινοειδή συμβάλλουν σε κάποιο βαθμό στα φαινόμενα αυτά. Αλλά αυτό δεν εμπίπτει ε, στην εντολή μας. Μελέτες παρακολούθησης, ναι. Έχουμε συλλέξει διάφορες ε, τέτοιες ε, μελέτες την ε, Μέλισσα, την μελέτη στην ε, Σλοβενία και αυτές έχουν ε, συζητηθεί αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης των επιρογνωμόνων μας. Αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε μια λυσίδα αιτιών ανάμεσα στο τι στα ευρήματα της μελέτης παρακολούθησης και τα νοικοτινοειδή. Τελικά δηλαδή δεν μπορέσαμε να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες από τις μελέτες παρακολούθησης. Ε, η προθεσμία ήταν πολύ σύντομη, ναι ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των συστάσεών μας. Ήταν ε, δύσκολο το να δουλέψουμε τόσο γρήγορα, αλλά ε, χρησιμοποίησαμε τους απαραίτητους πόρους και δεν πιστεύω ότι... Το χρονοδιάγραμμα είχε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την ποιότητα. Η ΕΦΣΑ ε, συνιστά να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Ναι. Και αυτό συνδέεται με μια από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη χρήση του εγγράφου καθοδήγησης που έχουμε ή της ε, επιστημονικής γνώμης που αποτέλεσε τη βάση για το έγγραφο αυτό. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη χρήση της επιστημονικής γνώμης ε, και ε, τα, τα, τα κενά δεδομένων ε, που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν. Ναι, πράγματι υπάρχει σχέση και γι' αυτό έχουμε καταγράψει μια σειρά κενών στα δεδομένα που θα θέλαμε να καλυφθούν για να έχουμε πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων των νεονικοτινοειδών στις μέλισσες. Κοιτώ τον κατάλογο των ερωτήσεων που τέθηκαν. Να συνοψίσω και πάλι κάποια στοιχεία κλειδιά των συμπερασμάτων μας. Ε, νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα νεονικοτινοειδή είναι πολύ τοξικά. Έχουμε τα δεδομένα σχετικά με την οξία τοξικότητα και τις μη θανατηφόρες ε, ε, επιπτώσεις είναι πολύ τοξικές οι ουσίες αυτές. Μελέτες ε, δείχνουν ότι έχουν ε, συμπεριφοριστικές ε, συνέπειες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορέσαμε να κάνουμε μελέτη, μελέτη σχετικά με τους κινδύνους. Σε κάποιες περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε ο κίνδυνος που υπάρχει. Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και Νομίζω ότι η έκθεση στη Σκόνη ή ε, στο νέκταρ και τη γύρι των ζαχαρότευτλων ε, ε, ή γενικά φυτών που δεν προσελκύουν τις μέλισσες σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε κάποιες μελέτες τις οποίες έχουμε μελετήσει. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ο κίνδυνος, σε άλλες περιπτώσεις όχι και δεν μπορούμε να καταλήξουμε με βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Στις περιπτώσεις αυτές ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αβεβαιότητα σε σχέση με, τις, ε, με την αξιολόγηση του κινδύνου που έχουμε κάνει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να έχουμε καλή κατανόηση του τι κάναμε, ποιοι είναι οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη δουλειά μας, που οφείλονται στην έλλειψη δεδομένων. Και αυτή ήταν η φιλοδοξία μας, να βεβαιωθούμε ότι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη έχουν κατανόηση του προβλήματος ε, και τώρα είναι εναπόκειται σε αυτούς να λάβουν ε, τις ε, σχετικές αποφάσεις. Εμείς προτείνουμε στην... Μάλλον η υποστήριξη που μπορούμε να παράσχουμε είναι οι περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη και οι κομισιόν δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα παράσχουμε τις πληροφορίες όπου είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων, εσά κύριε Χερμάν Φοντιέ, σημαντική ενημέρωση. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι μετά από αυτή την ευρεία συζήτηση είναι γεγονό ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι περαιτέρω έρευνε και μελέτε, διότι βεβαιότητε δεν διαθέτουμε. Πάντω, νομίζω θα επανέλθουμε και για αυτό το θέμα όταν ε, θα έρθει και ο Επίτροπος Μπόρκ. Θα ήθελα να περάσουμε αμέσω τώρα στο σημείο 4 της σημερινής διαταξής μας. Σημερινές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Είναι γνωμοδότηση του συναδέλφου του κυρίου Σπύρου Δανέλη. Αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατατέθησαν και τροπολογίες από τους συναδέλφους. Την περασμένη φορά δεν είχαμε χρόνο και αναβάλαμε την εξέταση του κειμένου για σήμερα και αύριο θα ψηφίσουμε. Και αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ήτρε Βιομηχανίας και Ενέργειας και θα λάβει υπόψη τη γνωμοδότησή μας για τη δική τους ψηφοφορία στις 18 Μαρτίου. Ε, δίνω το λόγο στο Σπύρο Δανέλη και συνάδελφοι να ζητήσουν από τη Γραμματεία. Αδελφοί, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το εξαιρετικό ενδιαφέρον σας για τη βελτίωση του κειμένου. Η γνωμοδότηση αυτή συντάχθηκε ξεκινώντας από τη διαπίστωση των συνθήκων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Γεωργία και τη σύνδεσή τους με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Οι σημερινές προκλήσεις λοιπόν είναι 1. Η κλιματική αλλαγή, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και η κατασπατάληση των φυσικών πόρων. 2. Η επισητιστική ασφάλεια, όσο και η ασφάλεια των τροφίμων. Τρία, Η αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας. Τέσσερα, Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, τηρώντας τις υποχρεώσεις έναντι του ΠΟΕ για την εξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. 5. Η αστάθεια στις αγορές γεωργικών προϊόντων, και έξι Η αποδυνάμωση των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της αδυναμίας αξιοποίησης συνεργειών από μεταξύ τους συνεργασίες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν και πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί η εξοικονόμηση της ενέργειας και η μείωση των απολειών ενέργειας και φυσικών πόρων. Οι δύο αυτοί στόχοι πρέπει να είναι αλληλοσυμπληρούμενοι και απόλυτα συνδεδεμένοι. Δεν αρκεί όμως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Στόχος μας δεν είναι μόνο η εξασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας υπό οποιοδήποτε κόστος. Στόχος μας είναι η βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της Ευρώπης, κατά τρόπο που να επιτρέπει την παράλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων που προανέφερα με τρόπο αποτελεσματικό. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο. Και αυτό έχει ήδη γίνει εμφανές στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, τα οποία είναι σε θέση να συμβάλλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής υπό τον όρο ότι θα έχουν ως τελικό καθαρό αποτέλεσμα πραγματική εξοικονόμηση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Ακόμη περισσότερο, οι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα δαπανηρό τρόπο μείωσης των εκπομπών που μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό θα πρέπει να αποτελεί και κομβικό στοιχείο στη χάραξη στρατηγικής και στην επιλογή μέτρων πολιτικής. Ο λόγος είναι ότι μια πολιτική μπορεί να εισάγει στρεβλώσεις που θα καταστήσουν τη φαινομενική ανταγωνιστικότητα μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Και αυτό μπορεί να έχει και κοινωνικές και οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για αυτούς τους λόγους υποστηρίζουμε ότι απαιτείται να δοθεί μεγάλο βάρος στην έρευνα και την καινοτομία και να αναπτυχθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι ενεργειακού εφοδιασμού από τους σημερινούς. Είναι με αυτούς τους τρόπους που θα μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε πραγματική και βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, καταπολεμώντας παράλληλα την κλιματική αλλαγή και προστατεύοντας φυσικούς πόρους και περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι συχνά είναι οι μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και διάδοση γνώσης. Ίσως η μεταβολή που μπορεί να επιφέρει αναμονάδα παραγωγής η καλύτερη κατάρτιση μιας μικρής εκμετάλλευσης να είναι μεγαλύτερη από τις δυνατότητες βελτίωσης που υπάρχουν με μεγάλες εκμεταλλεύσεις που συνήθως λειτουργούν με αξιοποίηση της τεχνολογίας κλίμακας. Γι' αυτό και θεωρούμε σημαντικό να προωθηθεί η γνώση για χρήση μικρής κλίμακας τεχνολογίας που εξοικονομεί ενέργεια χωρίς να απαιτεί μεγάλα έργα υποδομών και χωρίς να απειλεί τη βιοπικιλότητα ή να απαιτεί αλλαγές στη χρήση γης. Θα ήθελα τέλος να υπογραμμίσω τη σημασία που νομίζουμε ότι έχει η συνεργασία των αγροτών στο εγχείρημα διάδοσης των ενώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι βέβαιο ότι αν δεν πιστούν οι ίδιοι αγρότες για τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν, δεν θα πετύχουμε απόλυτη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Και για να υπάρχουν ωφέλη θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες οικονομίες κλίμακας που αποφέρει η συνεργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω ότι με αυτή την παρουσίαση να βοήθησαν να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους προτείνω την απόρριψη τροπολογιών συναδέλφων, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζω την προσπάθεια που κατέβαλαν για τη βελτίωση του κειμένου. Ελπίζω επίσης ότι έκανα σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε η συγκεκριμένη γνωμοδότηση και την οποία σας καλώ να υπερψηφίσετε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ Σπύρο. Και αμέσως αρχίζει η συζήτηση. Επτά συνάδελφοι έχουν εγγραφεί, αλλά προσοχή για να προκάνουμε. Γιατί θα έρθει ο Επίτροπος, η κυρία Ράιμερς και μετά η κυρία Γιούσο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Όλοι είμαστε υπέρ των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και πανευρωπαϊκά και καταρχήν. Αλλά από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει θέμα υπερεπιβάρησης και υπερφορολόγησης. Και δεν θα πρέπει μια στρεβλή εξέλιξη που γνωρίσαμε στη Γερμανία να γίνει ευρωπαϊκή. Προσοχή λοιπόν να μην βάλουμε πάρα πολλά χρήματα σε ένα κλάδο που τελικά μπορεί να είναι ανταγωνιστικός προς την παραγωγή τροφίμων και υπάρχουν και μεγάλες αντιστάσεις από τον πληθυσμό. Ε, έχουν ε, δοθεί μέτρα στήριξης που δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω τώρα γιατί έχει κάνει τον προγραμματισμό της η αγορά και υπάρχει και ένα ζήτημα υπερβολικής ε, καλλιέργειας αραβοσίτου. Μονοκαλλιέργεια σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, και πρόβλημα στη βιοπικιλότητα με ενδεχόμενες απώλειες εκεί. Αλλά ε, και επειδή φαίνεται αυτό και οπτικά σε μεγάλο βαθμό οι καλλιέργειες, έχει ε, ξεκινήσει μια αντίσταση ο πληθυσμός και θα πρέπει να κοιτάμε πού είναι τα όρια του εφικτού και κάποια στιγμή η ίδια η αγορά να αναλάβει και το κόστος. Και αν υπάρχει χρηματική ενίσχυση να είναι μια ε, κινητροδότηση για την έναρξη της δραστηριότητας και μετά αυτή να αυτονομηθεί και μπορεί να αυτοχρηματοδοτείται. Δεν μπορεί στο διηνικές να ε, επιδοτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουν να περπατάνε και μόνοι τους. Η κυρία Γιούσο και μετά ε, Άγνιο. Όχι κυρία Άγνιο, πρώτα η κυρία Γιούσο. Α, ζητώ συγγνώμη. Είναι τα ονόματά μας τόσο κοντά. Ε, κυρία Γιούσο, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας μιλήσω ε, ως σκιώδη συζητήτρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να συμφωνήσω με τη γνωμοδότηση του κυρίου Δανέλη στο σύνολό της σχεδόν και ήθελα να τον συγχαρώ κιόλα ε, για την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Ε, η ανακοίνηση αυτή δείχνει τους βασικούς τομείς που θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε οι ανανεώσιμες πηγές να φτάσουν ε, στους στόχους και να είναι και ανταγωνιστικές. Συμφωνώ απολύτως ότι έχει σημασία, όπως είπε η κυρία Ράιμερς, να μην είναι συνεχώς επιδοτούμενος αυτός ο κλάδος, αλλά να υπάρχει ένα δυναμικό χρειάζεται να τις βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους, μετά όμως να γίνουν ανταγωνιστικές ε, από μόνες τους. Να διευκολύνουμε αυτή τη μετάβαση ε, και να μπαίνουν στα δίκτυα ε, διανομής ενέργειας και καυσίμων από εκεί και πέρα. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, η βοήθεια για την πρόσβαση από τις ίδιες τις επιδοτήσεις. Έχω κάνει κάποιες τροπολογίες εγώ για Ανανεώσιμε πηγέ που έχουν ήδη λάβει σημαντικό βάρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν ένα ειδικό βάρο, το έχουν ήδη αποκτήσει από την πρώτη οδηγία που εγκρίθηκε πριν από μία δεκαετία και λίγο παραπάνω. Έχει αυξηθεί εντυπωσιακά ε, αυτό ο κλάδος έκτοτε στην Ευρώπη. Επίση, έχω και άλλη τροπολογία. Δεν είναι εναλλακτικέ πηγέ, άλλο είναι ανανεώσιμε είναι. Ε, στα ισπανικά, τουλάχιστον όταν λέμε εναλλακτικέ πηγέ είναι άλλο πράγμα. Και επίσης ε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα κριτήρια αηφορίας των βιοκαυσίμων υπάρχουν. Άλλο είναι αν θέλουμε να τα βελτιώσουμε, να τα αυξήσουμε, να τα αλλάξουμε. Υπάρχουν κριτήρια όμως ήδη αηφορίας και βιωσιμότητας. Και για μένα το σημαντικότερο είναι ε, να προωθηθούν τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς, γιατί έτσι θα γίνει φόρος και βιώσιμη παραγωγή και ε, δεν θα έχει επίπτωση στην παραγωγή τροφίμων το θέμα των καταλήπων και τη μείωσή τους. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε καλύτερη διαχείριση των πολυμάτων και των καταλήπων για να παράξουμε ε, προϊόντα και καύσιμα, βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Γενικά, συμφωνώ με όλες τις τροπολογίες, αλλά για την παράγραφο 7 οι τροπολογίες νομίζω δεν είναι καλές. Είναι καλύτερη διατύπωση του εισηγητού. Και Επίσης, διαφωνώ, μάλλον να το πω αλλιώς, συμφωνώ πολύ με την έρευνα. Και έχω κάνει και αντίστοιχη τροπολογία για τα βιοκαύσιμα ε, δεύτερης γενεάς. Αλλά όχι τα λεφτά από την αγροτική ανάπτυξη, είναι που είναι λίγα. Άμα τα βάλουμε και στην έρευνα για τις ανανεώσιμες, ε, νομίζω δεν θα γίνει καλή χρήση. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Αγνιού κύριος για ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Αγιούσο. Μιλάμε για προκλήσεις στον τομέα της γεωργίας με τις ανανεώσιμες και θα σας δώσω ε, μία πρόκληση. Ε, θα πρέπει να θέσουμε μία μεγάλη έκταση γεών ε, υπό μία ε, άλλη πηγή εναλλακτική για ανανεώσιμη, δηλαδή την ηλιακή ενέργεια. Αυτό αποτελεί μεγάλο σκάνδαλο και για μας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά επιδοτούνται και από τους φορολογούμενους οι οποίοι καταβάλουν το αντίτιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει στη δική μου ε, περιφέρεια Γκέρλινγκ και μετά Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Δεν έχουμε χρόνο. Με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα μαζί του. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι ύψης της σημασίας για τις ανανεώσιμες πηγές. Μιλάμε για μια ισορροπία μεταξύ αγροτικών προϊόντων, διατροφικής ασφάλειας και παραγωγής, καθώς και περιβάλλοντος. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα που φτάνουμε στην αναθεώρηση του κανονισμού της οδηγίας ε, για τις ανανεώσιμες και τη στιγμή που μιλάμε και για τη χρήση γεών άμεση και έμεση ή εναλλακτική, θα πρέπει να δούμε πού θα εντάξουμε και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας μέσα στα πλαίσια και των εξελίξεων στο γεωργικό τομέα. Η κυρία ε, Μαγκίνες δεν είναι εδώ, γι' αυτό το λόγο έχει ο Μάρτιν, Μάρτιν Μάρτιν, Μάρτιν Όσλιν. Μάρτιν και μετά ο κύριος Γκλάτενφέλτερ. Ναι, ε, επιγραμματικά μόνο για τη συζήτηση. Η κυρία Ράιμερ σωστά είπε ότι στη Γερμανία έχουμε ε, υπερβάλει αυτόν, ειδικά σε ό,τι αφορά τον αραβόσιτο και να μην πέσουν στα ίδια λάθη άλλα κράτη-μέλη. Ε, από τον υπερβολικό ζήλο ε, ε, να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλοιπα. Δεν τα χρησιμοποιούμε αρκετά για την ανακύκλωση και παραγωγή των εναλλακτικών καυσίμων. Δηλαδή ε, δεν ε, ε, υπάρχει η σύγκρουση μόνο μεταξύ τροφίμων και καυσίμων αλλά και τροφίμων ζωοτροφών και καυσίμων γιατί υπάρχουν και τα ζώα που πρέπει να ταΐσουμε και να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά χρειάζονται κίνητρα τα κράτη-μέλη γιατί σε αντίθεση με τον Άγγλο συνάδελφο πρέπει να πω ότι από την αηφόρο χρήση ενέργειας εποφελούνται και κάποιοι αγρότες αν μπορεί με την κοπριά να παράξει ε, βιοαέριο ένας αγρότης είναι ένα επιπλέον έσοδο αυτό. Για να πω κάτι τώρα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενεάς. Ε, από πλευράς Γερμανίας πρέπει να πω ότι πριν από χρόνια ε, να αποθέσαμε ε, πολλές ελπίδες ε, στο ξύλο ή στο άχυρο από τα κατάλοιπα να βγάλουμε καύσιμα. Αυτό εγκαταλείφθηκε γιατί δεν είναι κερδοφόρο και τελικά απεδείχθη αδιέξοδο. Ούτε έχουμε πια τόσο άχυρο που να το χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε καύσιμα. Ε, δεν θα πρέπει να βάλουμε εκεί πάρα πολύ ενέργεια. μόνο να επικεντρωθούμε στο φυτικό έλαιο. Είναι το μοναδικό καύσιμο που αξίζει πραγματικά. Ευχαριστώ. Γκλάτεν και μετά η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικέ και για τη γεωργία αλλά και για την αγροτική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα διότι ακριβώς εκεί μπορεί να παραχθεί το μεγαλύτερο ε, ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν δείτε τα σχέδια και των 27 κρατών μελών ε, για το πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέχρι το 2020 για τις ανανεώσιμες, θα διαπιστώσετε ότι ε, τα κράτη-μέλη προβλέπουν το μισό ε, να καλυφθεί από βιομάζα γεωργικής ή δασικής προέλευσης. Θα ήθελα να έρθω τώρα σε δύο τροπολογίες. Η μία είναι η μια ειναι παριθμόν 7 και έχω και μια άλλη τροπολογία που είναι η 49 την οποία έχουν συνυπογράψει και οι φιλελεύθεροι. Ε, αν δεν απατώμε, Τουλάχιστον έτσι άκουσα, δεν ξέρω αν κάνω λάθο. Οι σοσιαλιστέ θέλουν να τι απορρίψουν και τι δύο αυτέ τροπολογίε. Μα τι ζητούν οι τροπολογίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει και αυτή μια σειρά υποχρεωτικών στόχων, δεσμευτικών και υπολογισμένων ε, για ε, την περίοδο μετά το 2020. Μα γενικά οι σοσιαλιστές είναι υπέρ των ανανεώσιμων. Μα το σημαντικό θέμα σήμερα είναι υπάρχουν στόχοι και προοπτικές και μετά το 2020 για την περίοδο μετά το 2020 για να μπορούν να ε, γνωρίζουν ε, την απόδοση των επενδύσεων οι ενδιαφερόμενοι, για να μπορέσουν να προγραμματίσουν και τι θα γίνει την περίοδο μετά το 2020 και πώς θα αυξηθεί στο ενεργειακό μείγμα ε, η συμμετοχή των ανανεώσιμων. Ελπίζω τουλάχιστον μία από τις δύο αυτές τροπολογίες οι σοσιαλιστές να την υποστηρίξουν, γιατί μόνο έτσι θα αναπτυχθεί και θα ευδοκιμήσει αυτό ο κλάδο. Επίση να πω δύο λόγια και για την ηλιακή ενέργεια, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί πολύ συχνά ο κόσμος βάζει φωτοβολταϊκά σε ε, χωράφια. Ε, έτσι ακούγεται δηλαδή. Δεν ισχύει αυτό. Στην Ουγγαρία ε, οι αγρότες αντιτίθεται σε τέτοιου είδους ανάπτυξη εντός εισαγωγικών και δεν θέλουν να δώσουν εδάφη που είναι γόνιμα για την καλλιέργεια ή για τη δασοκομεία και δεν θέλουν να γίνουν χωράφια που θα σπέρνουν φωτοβολταϊκά και μάλιστα έτσι αλλάζει και η νομοθεσία αυτή τη στιγμή στην ε, Ουγγαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω την έκθεση αυτή. Θα ήθελα όμως να επιστέσω την προσοχή σας ε, και των Ευρωβουλευτών ε, ότι υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την βιοοικονομία που συμπεριλαμβάνει το θέμα αυτό. Και από ό,τι κατάλαβα δεν γνωμοδοτούμε στην ε, έκθεση αυτή, παρότι η βιοοικονομία έχει να κάνει με τη χρήση της φύσης, ε, του εδάφους ε, και της γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να θίξετε το θέμα αυτό και να δείτε γιατί δεν γνωμοδοτεί η Επιτροπή Άγκρη τη στιγμή που σχετίζεται με το θέμα που συζητάμε. Θα το Μαρία. Ζήτησα να ζήτησα να μιλήσω εξ ε, του συναδέλφου ο οποίο μόλις ήρθε, λέει ο κύριος ε, Γι' αυτό και θα του δώσω τη συναδέλφου. Γι' αυτό και θα τη δώσω το λόγο. Ε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Δανέλη για την εξαιρετική αυτή εργασία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλώς καταρτισμένη η έκθεση. Μίλησε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο και ως προς τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον. Έχουν μεγάλη σημασία για τις γεωργικές περιοχές και υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες για τους αγρότες να μειώσουν τα έξοδά τους ως προς τη θέρμανση και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την αυτάρκεια σε ε, ενέργεια που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν χρησιμοποιήσει σωστά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να γίνει ε, βιώσιμη χρήση ε, αν λάβουμε υπόψη και την ε, βιοποικιλότητα και τις κλιματικές αλλαγές, όπως πολύ σωστά τόνισε ο εισηγητής. Η πολιτική υπέρ της ενέργειας δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την επισητιστική ασφάλεια ή την ε, γεωργική ανταγωνιστικότητα. Και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της αποδοτικότητας της έρευνας στην ε, παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας, καθώς ε, και να δούμε και τα γεωργικά συστήματα, χρήση βιομάζας, καθώς και το ζωικό κεφάλαιο. Επειδή πρόκειται για ένα νέο και πολλά υποσχόμενα τομέα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας και αηφορίας της Επιτροπής σε σχέση με την, ε, τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και με βάση τη βιωσιμότητά τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την προϋπάρχουσα νομοθεσία και μία εποπτή όταν μιλάμε για κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα, θα πρέπει και τα βιοκαύσιμα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικολογική βιωσιμότητα μέσα στα πλαίσια και των οικονομικών και κοινωνικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη και την μείωση πηγών ενέργειας. Υποστηρίζουμε όμως αυτή τη γνωμοδότηση και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία. Ωραία, σας ευχαριστώ Κύριε Μάνερ. Δίνω το λόγο στον κύριο Δανέλη για σύντομα συμπεράσματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την επικοδομητική συμβολή ε, και κατά τη διάρκεια της ε, συνεργασίας μας με τους Χιώδης αλλά και στην υποβολή των ε, τροπολογιών όπως και στην αποψινή συζήτηση. Νομίζω ότι ε, συμφωνούμε όλοι ότι ε, στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Ε, το θέμα για το οποίο συζητάμε, όπως και απόψε αναφέρθηκε από συναδέλφους, έχει ήδη εμφανίσει στρεβλώσεις σε λανθασμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του. Ε, έτσι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ισορροπημένοι για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα και την οικονομική και την περιβαλλοντική και την κοινωνική βεβαίως. Όσον αφορά τις τροπολογίες ε, του συναδέλφου Gladfelder, ε, θέλω να πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να, έχουμε, να εστιάσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020. Θεωρούμε ότι σε αυτή την πορεία είναι υπερβολικό να ζητήσουμε ε, στόχους για την μετά το 20 περίοδο, ιδίως δε όταν ε, ζητάμε κατανομή των στόχων ανακράτως μέλος. Ε, θεωρούμε ότι είναι μαξιμαλιστικό και μας αφαιρεί την δυναμική των προσπαθειών μας. Γι' αυτό εστιάζουμε στον μέχρι το 20. Ε, τέλος θέλω να πω ότι βεβαίως νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η, η βιωσιμότητα δεν πρέπει να είναι φαινομενική ως προς τον ανταγωνισμό ε, με άλλες μορφές ενέργειας όταν υπάρχει η επιδότηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική βιωσιμότητα και μετά την πάροδο ε, της υποστήριξης με τους παρεμβατισμούς των επιδοτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δανέλη. Συνάδελφοι, το θέμα 5 της σας διάταξης αναβάλλεται. Γι' αυτό η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση απάτης θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνάντηση της Επίτροπης αλλά η υποβολή τροπολογιών ισχύει για τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο να καλωσορίσω καταρχήν τον Επίτροπο Τόνιο Μπόρς, που είναι υπεύθυνο για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, που θα μας μιλήσει για τις προσεχείς πρωτοβουλίες μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Υπάρχουν και θέματα ειδικού ενδιαφέροντος και επίκαιρου ενδιαφέροντος. Και εδώ μιλώ για το κρέας αλόγου σε προπαρασκευασμένα προϊόντα, καθώς και τα νεονικοτινοειδή και τις επιπτώσεις επί των μελισσών. Η ΕΦΣΑ μας έκανε μια παρουσίαση, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, και έγινε μια ανταλλαγή απόψεων που μας απασχόλησε όλους θα μας μιλήσετε και για την εφαρμογή της οδηγίας 2008-120 του Συμβουλίου για την προστασία των χείρων και χειροειδών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα, την εκτροφή των θηλαίων. Στη συνέχεια θα μιλήσουν οι συντονιστές και μετά όλοι οι συνάδελφοι. Ο Τόνιο Μπορς έχει τον ε, ο Τόνι Μπόζ έχει το λόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας, διότι ήταν πολλά θέματα, θέματα υποσυζήτηση, αλλά ήταν προσχεδιασμένα, ενώ άλλα όχι αλλά που έχουν προσλάβει νέα σημασία με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις. Θα ήθελα όμως να δούμε τι θα μας απασχολήσει μέχρι τώρα, ε, από τώρα μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Ε, οι επόμενοι 14 μήνες θα περάσουν τάχιστα και η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ύψης της σημασίας για να είμαστε αποδοτικοί. Ας αρχίσουμε με το θέμα το οποίο απασχόλησε τον τύπο τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή το κρέας αλόγου το οποίο υπάρχει σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε κράτη-μέλη. θα ήθελα να σταθώ σε δύο ή τρία σημεία. Καταρχήν, μέχρι τώρα αυτό το θέμα δεν ήταν ένα θέμα ασφάλειας τροφίμων. Ήταν θέμα σήμανσης προϊόντων κρέατος με απατηλό, απατηλή σήμανση για λόγους οικονομικού κέρδους αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ε, ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, δεν, πρόκειται για, δεν έχουμε ενδείξει ότι πρόκειται για κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται για θέμα έλλειψης ε, νομοθέτησης. Υπάρχει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σήμανση και αφορά τα προϊόντα κρέατος. Θα πρέπει δηλαδή ε, να έχουμε σήμανση για να ξέρουμε ε, τι προέλευσης είναι το ε, κρέας, ποιας προέλευσης δηλαδή. Το κρέας αλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η σωστή σήμανση. Επίσης υπάρχει το σύστημα της τάχης της ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και υπάρχει και η νομοθεσία σκοπιμότητας η οποία είναι και λειτουργική. Δηλαδή, μέσα σε μία-δύο μέρες μπορέσαμε να ανοιχνεύσουμε την προέλευση των προϊόντων ε, κρέατος και πού διήλθαν, από ποια κρατη δηλαδή. Και το δεύτερο... how αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, λανθασμένες αντιλήψεις, ότι δηλαδή η εφαρμογή της ε, κοινοτικής νομοθεσίας είναι βασικό μέλημα των κρατών μελών, που δεν σημαίνει βεβαίως ότι η Επίτροπη δεν ε, συντονίζει αυτές τις προσπάθειες και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα Αυτά τα τρία είναι τα τρία βασικά σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή δεν ε, ήταν αδρανής. Στις 13 ε, Φεβρουαρίου υπό Ιρλανδική Προεδρία έγινε μια έκτακτη συνάντηση υπό Ιρλανδική Προεδρία η οποία κατά τη διάρκεια της οποίας είπα ότι θα πρότεινα συγκεκριμένες δράσεις μέσα στα πλαίσια της ε, μόνιμης επιτροπής, η οποία και αποφάθηκε στις 15. Αυτή η πρόταση αφορούσε συγκεκριμένη εποπτεία που αφορούσε δύο στοιχεία. Μία σειρά δοκιμών DNA σε προϊόντα κρέατος, βοήου κρέατος, για να δούμε κατά πόσο ανοιχνεύεται ε, κρέας αλόγου. Of the absence of phenylbutazone, popularly known as in... Και θέλαμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει φενιλβουταζόνη στα, στο αλογίσιο κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες. Και έτσι έγινε μια σειρά δοκιμών και γίνεται μία ε, ε, σειρά δοκιμών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου για να δούμε κατά πόσο υπάρχει φενιλοβουταζόνη σε ορισμένα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το κρέας αλόγου όταν έχει ε, ενσταλλαχτεί από φενιλοβουταζόνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη χρήση. Και αυτό που μας ενδιέφερε είναι να δούμε ότι τη στιγμή που έχω έχει γίνει επεξεργασία κρέατος αλόγου με φενιλοβουταζόνη, δεν θα μπορούσε αυτό το κρέας να προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι δοκιμές αυτές θα διενεργηθούν για ένα μήνα με μία επιπρόσθετη περίοδο δύο μηνών. Ε, έγινε θετική γνωμοδότηση επ' αυτού και μέχρι τις 15 Μαρτίου η Επιτροπή θα γνωρίζει τα αποτελέσματα. Υπάρχει δέσμευση να δημοσιεύσουμε άμεσα αυτά τα αποτελέσματα. Όχι μόνο εξαιτία του ενδιαφέροντος που παρουσίασε αυτό το θέμα, αλλά και εξαιτία των ανησυχιών των καταναλωτών, έτσι ώστε να προωθήσουμε και τη μελλοντική μας δραστηριότητα με βάση τα αποτελέσματα αυτά. Ο αριθμός δοκιμών που θα διενεργηθεί σε κάθε κράτος μέλος θα είναι αναλογικός με το εμπόριο κρέατος, τον αριθμό των σφαγίων και, και, και ανάλογα με την ποσότητα του εισαγόμενου κρέατος αλόγου. Στη συνέχεια θα προβληθεί μια σύσταση όπως αποφάσισε η μόνιμη επιτροπή την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι, την 1η Μαρτίου θα εφαρμοστούν, θα διενεργηθούν οι πρώτες δοκιμές. Η Επιτροπή ενέκρινε αυτό το πρόγραμμα δοκιμών στις 19 Φεβρουαρίου και το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Όσο αφορά τις δοκιμές για την έλλειψη φενιλοβουταζόνης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρουμε ένα δείγμα 50 τόνων κρέατος ε, αλόγου, το οποίο έχει εισαχθεί με ένα ελάχιστο όρο 5 δειγμάτων ανακράτος μέλος. Η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει αυτό αυτούς, αυτές τις δοκιμές σε επίπεδο 75%. Δηλαδή θα καταβάλει 300 ευρώ αναδοκιμή. Τέλος, η Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 θα πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μία έκθεση για την σήμανση της προέλευσης του κρέατος που ε, χρησιμοποιήθηκε. Η προέλευση του κρέτος δεν έχει σχέση με αυτό το συμβάν. Εδώ είχαμε να κάνουμε με θέμα σήμανσης ως προς την προέλευση, ως προς την ε, προέλευση του κρέατος, δηλαδή κατά πόσο ήταν αλόγου ή όχι. Οι υπηρεσίες μου θα υποβάλουν αυτή την έκθεση πριν από το Δεκέμβριο και το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα θα ήθελα να στραφώ σε άλλα ζητήματα, δηλαδή να δούμε τις δαπάνες στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Έχει επιτευχθεί πρόοδος προς ε, μια συμφωνία μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, έτσι ώστε να δούμε πώς είναι η σωστή διαχείριση δαπανών σε σχέση με την αλυσίδα τροφίμων. Θεωρούμε ότι το προϋπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργεί καλώς και παρέχει πραγματική προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό δεν θα ζητήσουμε να επέλθει ρήξη ελευθή μεταρρύθμιση, απλώς να εξορθολογήσουμε το πλαίσιο για να είναι οι πολιτικές μας πιο αποτελεσματικές και να επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία. Υποθέτω ότι η πρόταση αυτή όταν δημοσιευθεί θα τύχει της αναγνώρισης και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και θα εγκριθεί αμελητή. Και τώρα φτάνω στην, ε, στις τέσσερις ε, τομεακές προτάσεις που αφορούν το πακέτο τροφίμων και ζωοτροφών και της ασφάλειάς τους. Χαίρομαι, ε, αλλά και λυπάμαι ιδιαίτερα διότι οι προετοιμασίες αυτές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Όμως οι προτάσεις αυτές θα εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν. Έτσι θα ενημερώσουμε, θα απλουστεύσουμε και θα διασαφηνίσουμε το τρέχον σύστημα το οποίο μας υπηρέτησε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να έχουμε πιο εστιασμένα μέσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους κινδύνους σε όλο το φάσμα της ε, διατροφικής αλυσίδας μιλώντας για την ε, υγεία των ζώων, των φυτών, των σπόρων και τους επίσημους ελέγχους. Επίσης ε, προβλέπεται αναθεώρηση του πακέτου υγιεινής τροφίμων. Θα πρόκειται για, μια, ε, για ένα εγχείρημα λεπτομεριών, καθορισμού λεπτομεριών. Τώρα, σε σχέση με την ε, ευημερία των ζώων. Of January of this year. Από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους ε, υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο για τους εκτροφείς και τις εκμεταλλεύσεις με 10 ε, ε, ε, χείρους και άνου. Και η θέση μας ήταν απόλυτα σαφής. Θέλουμε να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση σε όλα τα κράτη-μέλη για τους εκτροφείς χείρων και ιδιαιτερα φιλέων. φυλαίων. Δυστυχώς, ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, συμμορφωθεί πλήρως. Αύριο λοιπόν προβλέπεται με μία επιστολή η εκκίνηση των διαδικασιών παράβασης δυνάμει των συνθήκων. Τώρα, να στραφώ σε άλλα ζητήματα. Το Μάρτιο 2011 ε, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για τα, ως προς τα νέα, τις καινούργιες ζωοτροφές, τις νέες ζωοτροφές που αφορούν τις διατάξεις για την κλωνοποίηση των ζώων. Η Επιτροπή μετά από ευρύτατες διαβουλεύσεις και με βάση μία ακρόαση θα αποφανθεί τον Ιούλιο. Επίσης, ε, η πρόταση των νέων τροφίμων αντικατοπτρίζει τη Συνολική Συμφωνία του Μαρτίου 2011. Ας περάσω τώρα στις ε, μέλισσες και τη θνησιμότητα, τα νεονικοτινοειδή. Ελπίζω να μην ε, με κεντρήσετε ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αυτή. Αυτός ο κίνδυνος ε, εντοπίστηκε πρόσφατα, δηλαδή το ότι μπορούν να πληγούν οι μέλισσες από τη χρήση νεονικοτινοειδών. Αυτός ο κίνδυνος εντοπίστηκε από την ΕΦΣΑ. Θα ήθελα να πω ότι τους δυόμισι αυτούς μήνες της θητείας μου έχω ακούσει ότι η ΕΦΣΑ είναι ένα πολύ συντηρητικό όργανο, είναι ανέλικτο δεν έχει ιδιαίτερη ε, ευελιξία. Βλέπω όμως ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μελέτη που διενεργήθηκε ως προς τη χρήση των νέων που έχουν ε, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ε, μελισσών. Άρα δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να στυλιτεύω την ΕΦΣΑ τη στιγμή που αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την επιβεβαίωση αυτή, από την ΕΦΣΑ, το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, όπου πολλά κράτη-μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να λάβει τάχιστα και αναλογικά μέτρα. Θα ήθελα να ε, τονίσω ότι έχω λάβει μία επιστολή που έχουν συνυπογράψει 75 μέλη του Κοινοβουλίου ζητώντας από την Επιτροπή να απαγορεύσει τη χρήση όλων των νεονικοτινοειδών. Οι υπηρεσίες ε, της Επιτροπής άκουσαν εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη, έτσι θα μπορούσαμε να αναστείλουμε για δύο χρόνια τη χρήση των νέων οικοτινοειδών που έχει εντοπίσει η ΕΦΣΑ ότι δηλαδή αποτελούν πηγή κινδύνου. Έτσι αναγνωρίζουμε ότι σε μερικές ε, περιπτώσεις η ασφαλής χρήση αυτών των εντομοκτώνων είναι δυνατή. Και θα λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις αυτής της άμεσης δράσης στους ε, ενεχόμενους τομείς. Γι' αυτό μιλάμε για αναστολή για δύο χρόνια των ε, ε, τριών από τα έξι νεονικοτικονοειδών. Θα περιοριστούμε δηλαδή σε αυτά τα τρία ε, εντομοκτώνα στο σύνολο των έξι. Και μετά την ε, χρήση ε, τριών από αυτούς τους σπόρους μέχρι την πρώτη, μετά την 1η Ιουλίου 2013. Έτσι, τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν τη χρήση νεονικοτινοειδών σε σημαντικά, ε, σε σημαντικά είδη όπως τα ζαχαρότευτλα καθώς και τα σιτηρά κατά την περίοδο του χειμώνα. Και στη συνέχεια θα υποβληθούν ε, μέτρα, μάλλον θα υποβληθεί η έκθεση με μέτρα στη Μόνιμη Επιτροπή για γνωμοδότηση τον Μάρτιο. Είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα φιλόδοξα αποφασιστικά αλλά και αναλογικά μέτρα θα αντιμετωπίσουν, θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων, βελτιώνοντας την ε, υγεία των μελισσών επιτρέποντας παράλληλα στους αγρότες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εντομοκτάνα τη στιγμή που δεν ε, λοχεύει κίνδυνος. Παραμένοντας στο κεφάλαιο των μελισσών, και σε σχέση με τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο ως προς την οδηγία για το μέλι, θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση Επιτροπής δεν θα πρέπει να μεταλλαχθεί, να μετατραπεί σε ένα θέμα που να αφορά τους γενετικώς ε, τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Θεωρώ ότι ότι ε, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε το, το μέλι ως μεταποιημένο προϊόν, αλλά ως πρωτογενές προϊόν. Γιατί διαφορετικά οι καταναλωτές θα οδηγηθούν σε σύγχυση και δεν θα συμβαδίζαμε με τις διεθνείς προδιαγραφές. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αποφάσεις του ΔΕΚ η νομοθεσία περί γενετικώς ε, τροποποιημένων μηχανισμών θα ισχύσει και εάν βρεθεί μεταλλαγμένη γύρις στο μέλι, τότε θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως ισχύει και για άλλα προϊόντα, τη στιγμή που ανοιχνεύονται γενετικώς τροποποιημένες ουσίες. Αυτό αφορά ε, ένα μέτρο που ε, θα, εφησυχάσει, θα και τους ε, μελισσοκόμους και τους καταναλωτές. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχω καταφέρει να καλύψει όλο το φάσμα των θεμάτων που σας απασχολούν, αλλά πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα μπορέσετε να θίξετε οτιδήποτε θέμα, επιμέρους θέμα σας απασχολεί. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Επίτροπε για την πλήρη αυτή παρουσίαση του θέματος. Νομίζω ότι θα ανακύψουν πολλές ερωτήσεις και αρχίζουμε με τους συντονιστές. Μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στους συντονιστές και στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι υπόλοιποι βουλευτές που το επιθυμούν. Αλπερντές για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση ε, σχετικά με το επίκαιρο σκάνδαλο με το κρέας ύπου. Ε, συμφωνώ και σας υποστηρίζω. Το σύστημα ουσιαστικά λειτουργήσε, αλλά θα πρέπει να δούμε πού υπήρξαν ακόμα αδυναμίες. Λυπούμε ότι μόλις ε, υπάρξει ένα σκάνδαλο, πολλοί βγαίνουν και ζητούν νέα νομοθεσία και νέους κανονισμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν τα συστήματα και θα ήθελα να σας υποστηρίξω, να ελέγξετε, να ε, διαπιστώσετε κατά πόσο υπήρξαν κάποιες ε, ελλείψεις, κάποιες αδυναμίες για να ε, λυθούν και για επόμενα σκάνδαλα. Τι έχω ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν είναι αρμόδια βέβαια η Ευρώπη άμεσα. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη σε τέτοιες περιπτώσεις, για τέτοια εγκλήματα εντός εισαγωγικών, αν και δεν έχει αποδεχτεί και δεν μπορώ να το ισχυριστώ, θα πρέπει να υπάρχουν και ποινικέ κυρώσεις, όχι μόνο πρόστιμα, σε τέτοιες περιπτώσεις για να αποτρέπονται τέτοια ε, σκάνδαλα θα πρέπει να πίπτει και ράβδο στα κράτη-μέλη να αποφασίζονται ποινικέ κυρώσει ε, με φυλάκιση γιατί είναι εγκληματικέ ενέργειε και θα πρέπει να ε, ακολουθούν και οι απαραίτητες ποινικέ κυρώσεις. Ελπίζω τις επόμενες μέρες και εβδομάδες να ε, λυθεί αυτό το θέμα, να ε, αποκαλυφθεί όλο αυτό το σκάνδαλο με όλους τους ενεχομένους ε, που κρύβονται από πίσω. Υποστηρίζω και τα όσα είπατε μόλις για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Έχει και εδώ σημασία να είμαστε αντικειμενικοί και νυφάλιοι ε, ε, με προθεσμίες που να μπορούν να τηρούν και να προσαρμόζονται οι αγρότες αυτές. Σας υποστηρίζει πάρα πολύ η ομάδα μας τα όσα είπατε. Δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο από τους υπολείπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάπουλα Σάντος από τους Δημοκράτες. Ευχαριστώ και εγώ κατέγραψα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σε σχέση με την πρόσφατη ε, κρίση με τη σήμανση του κρέατος, δηλαδή ως προς τη λανθασμένη προέλευσή του και απατηλή σήμανση, διότι δεν πρόκειται για ε, κρέας αγελάδας, αλλά για κρέας λόγου. Πρόκειται για μία απάτη που ε, δεν είχε επιπτώσει στη δημόσια υγεία, αλλά δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες στους ε, καταναλωτές. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άλλοι οικονομικοί φορείς, οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι έντιμοι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει το σύστημα ελέγχου να είναι ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα των δεδομένων. Νομίζω ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να, είναι, να γίνονται, αν και γνωρίζω ότι πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δαπανηροί. Θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στους ελέγχους και να διαθέτουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα. Εντάχει, δύο-τρία ζητήματα θα ήθελα να θίξω. Μιλήσατε για μία νομοθεσία για την προέλευση του κρέατος και μιλάμε για την χρήση κλωνοποιημένων ζώων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα ήθελα να μας πει ο Επίτροπος ποια στρατηγική προβλέπει η Επιτροπή επί του θέματος. Τέλος, ως προς τους ε, γενετικώς τρεποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, θα υπάρχει σωστή ε, σήμανση, γιατί ακόμα και αν υπάρχουν υπολείμματα τέτοιων οργανισμών θα πρέπει να αναγράφονται στη ε, σήμανση. Ακόμα και αν πρόκειται για ε, αμελητές ποσότητες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές ε, επιχειρήσεις θέλουν να μετεγκατασταθούν εκτός Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες της ε, κοινή γνώμης χωρίς όμως να υπολοιπόμαστε ως προς τα μέτρα και τη στρατηγική που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επί του θέματος. George Lyon για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Μπορς στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Ήθελα να μας μιλήσει για κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Τρία βασικά θέματα θα ήθελα να θίξω, κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά το θέμα του κρέατος αλόγου. επικροτώ τις ε, δράσεις σας, παρότι κάποιοι λένε ότι έχουμε κλείσει την πόρτα ε, του, του στάβλου αφού τη δέσουμε το άλογο, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά που ε, αναγράφονται στην επισήμανση να είναι και αυτά που βρίσκονται μέσα στο προϊόν. Είναι πολύ σωστό το ότι ξεκαθαρίσατε ότι αυτό το θέμα δεν είναι θέμα ασφαλείας των τροφίμων, είναι θέμα εξαπάτησης του κοινού διότι νομίζουν ότι αγοράζουν ο κρέα και αγοράζουν αλογίσιο κρέας, το οποίο στοιχίζει το 1 τέταρτο της τιμή. Πιστεύω λοιπόν ότι σημαντικό είναι να βρούμε τους υπεύθυνους και να αναλάβουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να φροντίσουμε ε, οι υπεύθυνοι να διωχθούν για την εξαπάτηση του κοινού και ελπίζουμε η τυχαία δειγματοληψία να αποτρέψει τον κόσμο από το να ξαναπροσπαθήσει κάτι τέτοιο. Διότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι η επισήμανση, είναι το να διασφαλίσουμε η επισήμανση να συνάδει με το προϊόν. Επίσης, είπατε ότι 11 κράτη-μέλη συμμορφώνονται στην ε, απαγόρευση, αλλά ε, δεν μας είπατε τι γίνεται με τα 16 κράτη-μέλη που δεν ε, συμμορφώνονται με την ε, απαγόρευση. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που συμμορφώνονται κατά 99% ή κατά 60%. πότε θα μπορέσουμε να γνωρίζουμε ότι όλα τα προϊόντα στην Ευρώπη παράγονται νόμιμα, διότι υπάρχουν πολλά ε, προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά που έχουν ε, ε, παραχθεί παράνομα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχετε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη Άλλωστε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και τους παραγωγούς ε, που συμμορφώνονται τα τελευταία 9-10 χρόνια ε, έχοντας πληρώσει και το αντίστοιχο κόστος. Ε, τι θα κάνετε λοιπόν κατά των χωρών που δεν συμμορφώνονται, θα πρέπει να φροντίσετε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Και περνάω τώρα στα νεονικοτινοειδή. Ε, ανησυχούσα ότι η ανταπόκριση της Κομισιόν ε, είναι δυσανάλογη, διότι ε, φαινόταν σαν να προτείνετε εσείς απόλυτη απαγόρευση τα επόμενα δύο χρόνια. Εσείς είπατε τώρα στην παρουσίασή σας ότι θα γίνουν κάποιες εξαιρέσεις, μιλήσατε για τα ε, ζαχαρότεσλα, από ό,τι κατάλαβα ε, και οι χειμερινές ε, σπορές ε, θα εξαιρούνται. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ε, ποιε θα είναι όλες οι εξαιρέσεις. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση μιας ε, αναλογικής ανταπόκρισης, διότι η παρουσίαση που λάβαμε από την ΕΦΣΑ ε, ήταν πολύ ελλειπής όσον αφορά τα στοιχεία και δεν καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα. Φαινόταν να υπάρχει θεωρητικός κίνδυνος για τους πληθυσμούς μελισσών. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση που προτείνετε ώστε να είναι σαφές τι θέλετε να κάνετε δύο τελευταίες ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσετε. Ποια περιμένετε ότι θα είναι τα ωφέλη ε, του να εισαχθεί αυτή η απαγορεύση σε δύο χρόνια. Περιμένετε να δείτε αύξηση του πληθυσμού των μελισσών. Δεύτερον, ποιες ε, θα είναι οι ε, οι παρεμπίπτωσες επιπτώσεις της απαγόρευσης, διότι η ΕΦΣΑ σκεφτόταν την ε, έλεγε ότι η επιστροφή σε 9-10 διαφορετικά είδη εντομοκτώνων ε, για την καταπολέμηση της μελίγκρας ε, και των σαλιγκαριών θεωρούσε ότι είναι οπισθοδρόμηση. Μπορείτε να μας πείτε ε, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι συνέπειες και οι παρεπίπτουσες της απαγόρευσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Επίτροπο. Ε, οι ερμοδιότητές του καλύπτουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με την Επιτροπή μας και ελπίζω να μας επισκέφτεται συχνά διότι κάποια από τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όπως μόλις είπε ο κύριος Λάιον, ε, ε, ε, εξέφρασε κάποιες ανησυχίε. Θα ήθελα να σα θυμίσω κύριε Επίτροπε ότι πριν 14 μήνες ε, είχαμε ε, απαγόρευση στα κλουβιά και πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνονταν. Μα είπατε ότι αύριο θα στείλετε Ε, μας είπατε ότι θα ε, εκδώσετε σημείο μας σχετικά με την απαγόρευση ε, για ε, τα κλουβιά, αλλά είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, διότι πολλοί κτηνοτρόφοι πουλερικών σε όλη την Ευρώπη Υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι πουλερικών στην Ευρώπη. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό. Και όσον αφορά το θέμα του αλογίσιου κρέατος, ε, πολλά έχουν ήδη υποθεί και νομίζω ότι πολλά θα υποθούν και στο μέλλον, διότι υποψιάζομαι ότι η κατάσταση αυτή ε, δεν έχει τελειώσει καθόλου. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε ακόμα στο μέτωπο αυτό. Και θα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς ε, συνέβη. Μας ενδιαφέρει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, στα παραγόμενα προϊόντα. Έχω ακούσει αυτά που λένε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόβλημα ε, προτύπων των τροφίμων, είναι πρόβλημα εγκληματικότητας και συμφωνώ ε, διότι όπως είπε ο Τζόρτζ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι βρίσκεται στην επισήμανση βρίσκεται και μέσα στο πακέτο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε διάφορα πράγματα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και δεν είμαι ειδικό στο θέμα αυτό. Ε, υπάρχει αρκετός έλεγχος σχετικά με τη μεταφορά αλόγων. Και το ρωτώ αυτό διότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε. Ε, είδαμε πολύ ενδιαφέρον τους χάρτες που είδαμε στην τηλεόραση από την Πολωνία, στην Ολλανδία, στην Κύπρο, ε, παντού. Τι έλεγχο έχουμε ε, στους κρεοπόλες, τους χοντρέμπορους κρεάτων που κάθονται σε έναν υπολογιστή και αγοράζουν και πολλούν κρέας χωρίς να έρχονται σε καθόλου σε επαφή μαζί του. μάλλον θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το θέμα νομίζω ότι θα πρέπει ε, να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Πρόκειται για εγκληματική πράξη. Το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει και θα πρέπει να επιβάλλουμε σωστά τον νόμο. Επικροτώ αυτά που είπατε περί ε, δοκιμών DNA. Ε, αναφερθήκατε και στο θέμα του κόστους, αλλά κάποιος ε, θα πρέπει να πληρώσει. Και μακροπρόθεσμα θα πρέπει ε, ε, να εξετάσουμε τις συνέπειες. Ε, είδαμε το θέμα της σποκόδους κεφαλοπάθειας, του αυτόδους πυρετού. Δεν θέλω να ξαναδώ τέτοιες καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και πόσο μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα και να αφήνουμε τους ε, λιανεμπόρους να ε, κατηγορούν τους ε, χοντρέμπορους και τους παραγωγούς. Και αυτοί οι λιανοπόλες έχουν ευθύνη, πιστεύω, και θα πρέπει και αυτοί να πληρώσουν το τίμημα. Έχω πολύ ισχυρές γνώμες για το θέμα αυτό και νομίζω ότι και εσείς το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι καταναλωτές στα κράτη-μέλη μας και σε όλη την Ευρώπη να γνωρίζουν τι αγοράζουν, διότι μπορεί ε, στην περίπτωση αυτή να μιλάμε για μικρό αριθμό ανθρώπων, ε, ε, αν κοιτάξουμε το σύνολο του τομέα αυτού, αλλά καταστρέφουν τις συνθήκες για τους άλλους που είναι νομοταγής και ακολουθούν τους κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρτιν Χόισλινγκ. Ναι. Χαίρομαι κύριε Μπορς που είστε εδώ. Μακάρι να ερχόσασταν συχνότερα. Γιατί σίγουρα χρειάζεται εκτενέστερη συζήτηση από όσο μπορούμε σήμερα να διευκρινίσουμε. Θα έρθω και εγώ στο σκάνδαλο με το ήπιο κρέας. Εξεπλάγει από αυτά που άκουσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι ορίστε αυτό είναι απόδειξη ότι όλα πάνε ρολόι στην Ευρώπη επειδή τώρα το ανακαλύψαμε. Μα το αντίθετο συμβαίνει. Δεν το ανακάλυψαν οι αρμόδιες αρχές και τώρα είμαστε τέσσερις εβδομάδες μετά το πρώτο έβριμα και ακόμα εξακολουθεί να ανοιχνεύεται ήπιο κρέας ε, με ε. Και ποιος ξέρει είναι το τελευταίο. Και ένα ε, πρόβλημα που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε καλύτερη ίχνη λασιμότητα, το απέρριψε ο, Συμβούλιο Υπουργό. Τώρα εσείς θα πρέπει να καταθέσετε ε, μία έκθεση ε, κάντε το νωρίτερα από το φθινόπωρο για να γίνεται καλύτερη και η καταγραφή και η αναφορά των κρεάτων. Ξέρω πάντα θα υπάρχουν κάποιοι εγκληματίε, αλλά ε, θα πρέπει να βρούμε πιο γρήγορα τους κρίκους της αλυσίδας. Και ο Τζιμ είπε κάτι και έχει απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν έμποροι και ξανάρχονται και δραστηριοποιούνται ως ε, έμποροι. Ε, δεν υπάρχει καμιά μαύρη λίστα. Πολύ περισσότερο κρέας που εισάγεται από ό,τι δηλώνεται. Και τελικά κλονίζεται ή χάνεται για η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Άλλο ένα σκάνδαλο. Και στην αρχή μήπως προσπαθήσατε να το υποτιμήσετε ότι δεν είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας και προστασίας του καταναλωτού, ότι ήταν απλώς απάτη. Ε, ε, ε προσπαθήσατε λίγο να ρίξετε τους τόνους. Και τι γίνεται με τους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Τα παίρνει σοβαρά όλα αυτά υπόψη τη συνένωση να υπάρχει ε, ενιαίος έλεγχος ο ίδιος όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται επιτέλους ε, το ίδιο επίπεδο για να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύουν παντού τα ίδια. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω. Αναφερθήκατε στη γενετική τεχνολογία έτσι μόλις ακροθυγός. Ε, γίνεται τώρα συζήτηση για την επανεθνικοποίηση της αδειοδότησης. Δεν έχει λυθεί το θέμα πώς θα προχωρήσετε. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι μέχρι να υπάρξει νέα ρύθμιση δεν θα έχουμε και νέα έγκριση για γενετικά τροποποιημένα φυτά. Γιατί μας προβληματίζει αυτό και η μηδενική ανοχή ήρθε αυτή η μηθενική ανοχή για τις ζωοτροφές. Ρωτήσαμε τις υπηρεσίες σας και... Δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα ε, στις ζωοτροφές. Γιατί ήρθε λοιπόν αυτό το μέτρο, καταργήθηκε η μηδενική ανοχή στις ζωοτροφέ. και για τα τρόφιμα θα κάνετε το ίδιο, γιατί αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, για την κλωνοποίηση, μια τελευταία ερώτηση. Και στην ακρόαση σα είπατε ότι θέλετε ταχεία λύση, αλλά τώρα δεν είπατε ποια λύση θα είναι αυτή. Τι γίνεται και με την επόμενη γενεά. Δηλαδή, έχουμε ένα κλωνοποιημένο ζώο οι απόγονοι του θα ε, επισημαίνονται επίση. θα ξέρουμε ότι ε, προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Και ένα τελευταίο. Για ε, αλλαγή και κατεξαίρεση συμφωνούμε με τους επένους που απευθύνατε προς την ΕΦΣΑ για τα νέο νοικοτινοειδή. Ελπίζω να δοθεί συνέχεια στη μελέτη της ΕΦΣΑ. Χρειάζεται βέβαια και άλλη διερεύνηση, αλλά δεν μπορούμε παρά να την υποστηρίξουμε. Είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση να απαγορευτούν πλήρως τελικά αυτές οι ουσίες. Ευχαριστώ Μάρτιν. Ο κύριος Μπλουμ από την Ομάδα της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Έκανα μια ομιλία του 2009 για το αλογίσιο κρέας, όπου εξέφρασα κάποιες από τις ανησυχίες μου σχετικά με τη συγκεκριμένη πτυχή. Επίσης ε, θυμάμαι ότι πριν 10-12 χρόνια μιλούσα για την εξαφάνιση των ε, Βρετανικών ε, σφαγίων τότε που έκλεισαν ε, χίλια σφαγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων. Με όλα τα προβλήματα που αυτό σήμαινε για την ε, ευζοία των ζώων, την υγιεινή του κρέατος και διάφορα άλλα πράγματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο κόσμο των καταναλωτών. Με 27 διαφορετικές χώρες, ε, με διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, Φαίνεται να μην υπάρχει φρένο στο τι μπαίνει στο φαΐ και ε, το τι σημαίνει ευσοία. Ε, θα συμφωνήσω με τον Τζιμ Νίκολσον ε, ότι το πρόβλημα εδώ είναι της επιβολής του νόμου. Ο Τζιμ Νίκολσον πολύ σωστά αναφέρει το θέμα της εφαρμογής των κανόνων και δεν ξέρω ε, αν ε, μπορούν να το μεταφράσουν αυτό οι διερμηνείς, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια λύση τύπου Χιθ ε, Είναι πάρα πολύ δύσκολο 27 κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και να συμμορφωθούν και εγώ θα υποστήριζα ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση όπου, το, ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει άλλη μία αρμοδιότητα αλλά επιδεικνύει ανικανότητα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αρμοδιότητα θα πρέπει να επιστραφεί στα κράτη-μέλη που μπορούν να ε, εφαρμόσουν τα πράγματα αυτά πολύ καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κάτι τέτοιο φαίνεται να συνειδητοποιεί σιγά σιγά και το Βρετανικό κοινό. Ευχαριστώ. Ρουμπίξ, τελευταίο συντονιστή από πλευρά των κομμουνιστών, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Χαίρομαι και εγώ κύριε Επίτροπε που σας λέω στην Επιτροπή μας και ε, πήρατε θέση ε, όχι μόνο για αυτό το σοβαρό ζήτημα αλλά και για άλλα θέματα πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, την αρχική σας τοποθέτηση και το ερμηνεύω ως εξής. Ε, ότι η νομοθεσία είναι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συνεχίζουμε τις δοκιμές. Μα αν είναι εντάξει η νομοθεσία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τότε μήπως δεν είναι έλεγχη. Έχουμε αρκετούς ελέγχους. Έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους, αν είναι σωστή η νομοθεσία. Βέβαια θα σου πει όλος ότι δεν μπορούν να τα ελέγχουν πάντα ε, οι Ευρωπαίοι ελεγκτέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά ζητήσουμε επιθεωρήσει τότε από τα κράτη-μέλη. Γιατί βλέπουμε διάφορες ασθένειε. Πότε αρρωσταίνουν τα πουλερικά, πότε αρρωσταίνουν οι χείροι, πότε έχουμε προβλήματα με ε, αλογίσιο κρέας. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να ε, σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα επισήμαση. Βασικά είναι αξιόπινη πράξη, απάτη. Εδώ και ένα μήνα το συζητάμε και ακούμε διάφορα. Συμπέρασμα κανένα όμως. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να λύνουμε τα πάντα με την νομοθεσία και με την ε, σωστή υλοποίησή της. Χαιρετίζω τους ενισχυμένους ελέγχους που αναφέρετε κι εσείς. Δεν ξέρουμε πού ήταν το πρόβλημα. Μπορεί κατά την πώληση να δηλώθηκε ότι ήταν κρέας αλόγου και τελικά να χάθηκε αυτή η αναγραφή κατά την επεξεργασία του κρέατος δεν ξέρω που έγινε. Πάντως έχουμε αποφασίσει εμείς πολλές ρυθμίσεις, πολλούς νόμους. Από ό,τι φαίνεται παραθυράκια υπάρχουν πάντα. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν είχατε την ευκαιρία να ελέγξετε αυτά τα παραθυράκια στην νομοθεσία και στην εφαρμογή της. Και τι πταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι πολύ χαμηλές οι απαιτήσει μας από τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους για να προχωρήσουμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συντονιστές. Ως ήθιστε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στους συντονιστές και μετά θα παρέμβουν και οι άλλοι συνάδελφοι γιατί έχουμε 20 εγγεγραμμένους. Ο Τόνιο Μπόρς έχει το λόγο, ο Επίτροπος. Ε, εκτίμησα ε, ιδιαίτερα τη μεταφορά ε, του κυρίου λάιν δηλαδή το λογοπαίγνιο που έκανε σε σχέση με το κρέας αλόγου, δηλαδή ότι δράσαμε αφού αγοράστηκε το άλογο. Έχουμε μια εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, μιλάμε για μεταφορά αγαθών, ε, υπάρχει η νομοθεσία, δεν υπάρχει θέμα έλλειψης ε, νομοθέτησης και όπου υπάρχει νόμος υπάρχει και ο παραβάτης του. Το οποίο δεν σημαίνει ότι ο νόμος ε, δεν είναι καλός ή ότι δεν υπάρχει σωστή θέση σε ισχύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το ανακάλυψε ένα κράτος μέλος, δηλαδή ένας οργανισμός τροφίμων στην Ιρλανδία ε, εξετάζοντας τα χάμπερκερ είδε ότι μέσα στο περιεχόμενο υπήρχε και κρέας αλόγου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε νομοθεσία σε ισχύ σε ένα κράτος μέλος το οποίο οδήγησε σε μια αυστηρή εποπτεία όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε ε, κρίση, όχι μόνο σε αυτή που αφορά την επισητιστική αλυσίδα, την αλυσίδα τροφίμων. Άρα το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να καταλύσουμε την εσωτερική αγορά και να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να επαναφέρουν απαγορεύσεις όπως το κρίνουν για θέματα που δεν είναι θέματα ασφάλειας τροφίμων. Εδώ μιλάμε για μία απατηλή σήμανση. Και η απατηλή σήμανση δεν είναι θέμα ασφάλειας ε, τροφίμων. Δεν ε, ε, υποβαθμίζω αυτή την απάτη ή την παραβίαση του νόμου, αλλά είχαμε άλλα ζητήματα στο παρελθόν που οδήγησαν σε κινδύνους ως προς την ασφάλεια τροφίμων και παρεμφερείς κρίσης. Γι' αυτό κανένας δεν υποβαθμίζει και κανένας ε, δεν ακυρώνει τα πλεονεκτήματα του να υπάρχει μια πραγματικά εσωτερική αγορά, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μετακίνηση αγαθών ή προϊόντων, δεν θα πρέπει να είμαστε και προκατηλημένοι ως προς την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένες χώρες, γιατί εγώ όταν ανέκυψε η κρίση δεν κατονόμασα καμία ε, χώρα και η εταιρεία Beef Lasagna θα μπορούσε να θεωρηθεί υπέτεια. Αλλά εγώ έκρινα πρώτα ότι θα πρέπει να ε, γίνει έρευνα και ορισμένα κράτη-μέλη όρισαν και κατονόμασαν τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν εμπλεκόμενες. Θα μπορούσα να σας αναφερθώ σε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία μας κοινοποιήθηκαν. Όπου βλέπουμε ότι υπήρχε μία σειρά κρατών που έλαβε, παρέλαβε προϊόντα από αυτή την γαλλική εταιρεία, τη γαλλική επιχείρηση, 19 ήταν αυτές, τρεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπόλοιπες εντός, όπου ανιχνεύθηκε κρέας αλόγου από μία ε, συγκεκριμένη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, και είχαμε και κοινοποιήσεις με βάση το σύστημα ε, ταχείας ε, επισήμανσης σε σχέση με την παρουσία κρέατος αλόγου σε τέσσερις χώρες. Είχαμε έξι κοινοποίησης λοιπόν σε τέσσερις χώρες και αυτή τη στιγμή διενεργούνται ανακρίσεις. Τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, εκτός από τον τομέα του περιβάλλοντος, δεν ε, επιβάλλει ε, κυρώσεις. Δηλαδή δεν αναφέρεται άμεσα σε κυρώσεις, αλλά υπάρχει η τακτή διάταξη η οποία αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιβάλλουν τις κατάλληλες ποινές χρηματικές ινή, έτσι ώστε ε, να προβάλλουμε συγκεκριμένες κυρώσεις αποτρεπτικού χαρακτήρα. Και βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προβάλλουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Κάποιο μπορεί να την προβάλλει, άρα καταλαβαίνετε ότι πάντα φαινόμαστε χαμένοι. Εν πάση περιπτώσει, με βάση και την αρχή της επικουρικότητας μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μέσα σε ορισμένες παραμέτρους. Και νομίζω ότι οι ποινικέ κυρώσει είναι επαρκείς για να αναχαιτήσουν μελλοντικά τέτοια συμβάντα αλλά υπάρχει ας πούμε νόμος κατά των διαρρήξεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν διαρρήξεις στα σπίτια μας στο μέλλον. Δεν μπορώ να σας δώσω εγγυήσεις και να σας πω ότι τώρα, εδώ και τώρα, από, τις, ε, από τα εκατοντάδες ή χιλιάδες νομοθετήματα δεν υπάρχει κάποιος τώρα ο οποίος ε, παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συμβάν για να υποσκάψουμε την ε, εμπιστοσύνη που έχει ο καταναλωτής στο σύστημά μας ως προς την ε, διατροφική ασφάλεια, εντός και εκτός Ευρώπης. Εάν το ζήτημα αυτό που δεν είναι θέμα επισητιστικής ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, θεωρηθεί ως ε, τέτοιο, τότε παίρνει άλλες διαστάσεις. Στο παρελθόν είχαμε τέτοιες κρίσης ε, ε, και ως την, ε, όπως ίσχυσε και με την περίπτωση της τρελής αγελάδας που σε μία χώρα είχε επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις που ανέρχονταν στο 1% του ΑΕΠ Θα πρέπει λοιπόν να καταγράφουμε τα γεγονότα όσα έχουν, να μην υπερβάλλουμε, να μην τα διονγκώνουμε, αλλά να αποστέλουμε ένα μήνυμα λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις καλύτερες περιφέρειες του κόσμου, ε, ζώνες ε, του κόσμου ως προς την ασφάλεια τροφίμων και ότι το θέμα αφορά καθαρά ένα ζήτημα σήμανσης, απατηλής σήμανσης. Θα μεριμνήσουμε ώστε να μην επαναληφθεί γνωρίζοντας ότι επειδή υπάρχει μία εσωτερική αγορά υπάρχουν ε, προϊόντα κρέατος τα οποία περνάνε τα σύνορα και πάνε από τη μία χώρα στην άλλη. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να έχουμε αυστηρότερη νομοθεσία περί σήμανσης, είπα ότι ήδη αυτό το εξετάζουμε. Περιμένουμε την ε, έκθεση για την σήμανση σε σχέση με την προέλευση των προϊόντων αυτών. Δηλαδή όταν ε, λέμε για ε, προέλευση, όταν μιλάμε για προέλευση πολλές φορές ας πούμε για ένα παιχνίδι δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση. Μιλάμε για, για το αρχικό υλικό, για το μεταποιημένο προϊόν και ούτω καθεξής. Βάση περιπτώσει αναμένουμε αυτή την έκθεση και μετά θα αποφανθούμε ως και προς ε, θέματα σήμανσης. Βεβαίως υπάρχουν παραθυράκια και κενά στη νομοθεσία και στην θέση σε ισχύ του νόμου. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά ακόμα και με τη σωστή ισχύ ενός νόμου δεν μπορούμε να έχουμε τέλεια εφαρμογή ολόκληρου του νομοθετικού πλαισίου παντού, παντού και πάντα. Ως προς άλλα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν, πέρα από το κρέας λόγου, ας μιλήσω για τη διαδικασία ε, ε, παραβίασης για, ως προς την οδηγία για τις οτόκες όρνηθες έχει ληφθεί, ε, έχει αναλυφθεί η δράση και ε, μόνο δύο κράτη-μέλη σήμερα δεν ε, έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία περί οτόκων και νομίζω ότι προβλέπεται, συγκεκριμένα προβλέπονται κυρώσεις σε σχέση με τις, εγγύ, με τις 90% νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε για συμμόρφωση. Υπάρχουν δύο-τρία κράτη-μέλη όπου η συμμόρφωση ανέρχεται σε ένα 73-74%. Ε, έχουμε όμως και χώρες που συμμορφούνται σχεδόν ε, πλήρως. Και αυτό βεβαίως δεν συνάδει και με τον, ε, τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Και γι' αυτό θα γίνουν οι προσφυγές, οι προσφυγές που απαιτούνται έτσι ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή συμμόρφωση. Μετά από μία τόσο μακρά μεταβατική περίοδο που είχαμε, κλωνοποίηση. Προτίθεμε να απαγορεύσω, η Επιτροπή θα απαγορεύσει την εισαγωγή κλωνοποιημένων ζώων στην ε, αλυσίδα τροφίμων. Αυτό έχει ε, συζητηθεί και στο μέλλον και εδώ ε, μιλάμε και για νεοσούς που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο μηχανισμός ανιχνευσιμότητας έτσι ώστε να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο ως προς το γενετικό τροποποιημένα για τις ζωοτροφές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει εναρμονισμένη ανιχνευσιμότητα έτσι ώστε οι δοκιμές και οι έλεγχοι να γίνονται κατά εναρμονισμένο τρόπο. Θα προβάλλω, θα προωθήσω την σχετική ε, πρόταση νομοθετήματος και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη να τη θεωρήσουν λογική. Γιατί βασίζεται στην επικουρικότητα, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ε, με βάση μια αιτιολογία που ε, έχει να κάνει με άλλους τομείς πέρα από του περιβάλλοντος, γιατί το περιβάλλον δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Κομισιόν, δηλαδή να βασιστούν σε λόγους ασφάλειας ε, τροφίμων και να και έτσι θα προωθήσω και αυτή την πρόταση ε, σχετικά με τις καλλιέργειες με, γενετικός, ε, με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Α, με συγχωρείτε, ξέχασα το θέμα των μελισσών. Η πρόταση είναι αναλογική, επειδή περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα στοιχεία τα οποία η ΕΦΣΑ έχει ανοιχνεύσει ως ε, επικίνδυνα. Πρόκειται για μία απαγόρευση για την επεξεργασία σπόρων ε, και καλλιεργιών ε, που προσελκύουν τις μέλισσες δεν θα λάβουμε υπόψη το, τα κλειστά περιβάλλοντα ή τα φυτόρια, αλλά είμαι επιδεκτικό σε προτάσεις από τα κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα μέτρα, έτσι ώστε το θέμα αυτό να καταστεί ακόμα ε, περισσότερο αναλογικό. Ξέρω ότι το θέμα αυτό οδηγεί σε διχογνωμίες, Υπάρχουν εναλλακτικές ως προσορισμένα εντομοκτώνα τα οποία επιτρέπονται υπό συνθήκες, έτσι ώστε να αποφύγουμε αρνητικές συνέπειες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Νομίζω ότι με τη δεύτερη παρέμβασή σας έχουν διασαφινιστεί πολλά και έτσι ελπίζω ο μακρύς κατάλογος των ομιλητών να επιβραχυνθεί κάπως. Μιλάμε για 20 ομιλητές μέσα σε 20 λεπτά. Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε πολύ συνοπτικοί. Ένα λεπτό έχετε όλοι. Μαγκίνες καταρχήν. Thank you. Rather than a question... Ευχαριστώ. Ερώτηση. Μάλλον αντί να ρωτήσω, θα ήθελα να πω στον ε, Επίτροπο ότι νομίζω κινδυνεύουμε να ε, ε, θεραπεύουμε τα συμπτώματα αλλά όχι τις αιτίε. στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι να έχουμε δίκες και πιο ε, βιώσιμες σχέσεις στην αλυσίδα ε, παροχής τροφίμων. Είπαμε ότι ναι, πρόκειται για έγκλημα, πρόκειται για εξαπάτηση κατά την επισήμανση. Έχουμε σπασμένη αλυσίδα παροχής τροφίμων. Νομίζω λοιπόν ε, ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή και νομίζω ότι φοβόμαστε να ε, πειράξουμε το θέμα αυτό ε, επειδή φοβόμαστε να παρέμβουμε στην αγορά. Αλλά ε, υπάρχει πρόβλημα στην αγορά και η Επιτροπή Γεωργίας και η Επιτροπή Περιβάλλοντος είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε την κατάσταση, να φροντίσουμε η αλυσίδα παροχής τροφίμων να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Άλβες, θα ήθελα να μιλήσω ως προς το θέμα της οδηγίας περί καπνού. Το, ένα, το 50% της εξωτερικής επιφάνειας του κουτιού θα πρέπει να φέρεται σε ολέθριες συνέπειες επί της υγείας. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτή τη διάσταση που σας δείχνω. Πιστεύω ότι η ελάχιστη επιφάνεια σημαίνει ότι παίρνουμε το ίμιση και πάνω. Ε, στη δική μου περιοχή έχουμε δύο ε, εργοστάσια που καλύπτουν το 50% της αγοράς και εάν επιβληθεί κάτι τέτοιο της, ε, ως ελάχιστη προδιαγραφή θα υπάρχουν συνέπειες δηλαδή διατρέχουμε κίνδυνο και μπορούν να χάσουν αυτοί οι άνθρωποι την εργασία τους γιατί ε, αυτές είναι οι διαστάσεις των δικών μας πακέτων και όχι οι γνωστές που γνωρίζετε, οι τυποποιημένες. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Υποστηρίζω πολύ το όσα υπόθηκαν για το θέμα της τροφικής αλυσίδας. Είναι κεντρικό αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να μειωθεί να, το μέγεθος της να βραχύνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δύο πράγματα ακόμα συγκεκριμένα για τη διατροφή. Τα ε, ζωικά αλευρά έχουν επανεισαχθεί στην αρχή για τη διατροφή των νυχθείων και μετά ε, των ε, πουλερικών και των χείρων. Είναι τρομερή καταστροφή και τώρα που έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Λοιπόν, είτε θα αναθεωρήσετε αυτή σας την απόφαση, είτε για τους καταναλωτές, επαναλαμβάνω, είτε θα αναθεωρήσετε αυτή την έγκριση, είτε θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει ετικέτα για να γνωρίζουν οι καταναλωτές αν χρησιμοποιήθηκαν ζωικά άλευρα για τη διατροφή των ε, ψαριών και μετά των πουλερικών και των χείρων. Ε, τελευταία απόφαση που ελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου ε, είναι πάλι ένα ζήτημα εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές. Στις 4 Φεβρουαρίου υπογράψατε μία εκτελεστική απόφαση για να πείτε ότι για την τρελή αγελάδα, ε, για τα βοηδή, για τις αγελάδες συγκεκριμένα ηλικία άνω των 6 ετών. Τέτοιε ώρες, τέτοια λόγια. Να λέμε ότι θα σταματήσουμε οι δοκιμές και θα επιλέγουν τα κράτη να τις σταματήσουν. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ακόμα και αν 28 ε, μόνο ζώα ε, βρέθηκαν φέτος, είναι 28 ζώα που δεν έπρεπε να είχαν κυκλοφορήσει. Παρακαλώ να αναθεωρήσετε αυτή την απόφαση διότι οδηγεί σε σύγχυση τους καταναλωτές αλλά τελικά και τους κτηνοτρόφους γιατί σε τελική ανάλυση πάντα την ύφη την πληρώνει ο κτηνοτρόφος. Ένα τελευταίο. Ε, ε, στις νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, στις 25 Φεβρουαρίου θα μιλήσετε για τα μεταλλαγμένα θα κάνετε μελέτες για τις νέες ε, διεδοτήσεις και για τις παλιές εγκρίσεις θα γίνουν οι δοκιμές. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Συγγνώμη για την ταχύτητα και τους διερμηνείς. Ζητώ συγγνώμη. Αλγουάρτ και μετά η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος και θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, κοινέ έρευνες ε, Europol Interpol για τις ε, απάτες στα τρόφιμα. Η έρευνα αυτή είναι σχετικά πρόσφατη. Ε, κύριε Πίτροπε, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ε, η Ιρλανδική Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων βρήκε την απάτη αυτή και η έκθεση αυτή και άλλες εκθέσεις έδειξαν ότι οι έρευνες DNA έγιναν στην Ιρλανδία. Με εξέπληξε το ότι αυτό δεν αποτέλεσε αφορμή για την Κομισιόν τότε να αυξήσει την επαγρύπνηση όσον αφορά την απάτη στα τρόφιμα. Επιπλέον, έχω θίξει το θέμα αυτό στο γραφείο σας ε, το 2012 ε, με μια κοινοβουλευτική ερώτηση και στην απάντησή σας με ενημερώσατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έβλεπε την ανάγκη να αναπτύξει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης ε, στα τρόφιμα. Δηλαδή, εσείς είχατε φυσικαστεί παρότι είδαμε να χτυπάνε αγερμή σε όλη την Ευρώπη. Τώρα όμως βλέπουμε ότι το σκάνδαλο με το κρέας επηρεάζει όλο και περισσότερο περισσότερους πολίτες στην Ευρώπη, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και ε, εκατομμύρια ε, ευρώ. Ε, και βλέπουμε ότι παρά ήταν χαλαρή η στάση της Κομισιόν και διακυβεύει έτσι τους καταναλωτές και την βιομηχανία τροφίμων. Έχουμε συνέχεια ελέγχου ε, στι ε, αγροτικέ εκμεταλλεύσει, αλλά ε, κάτω από τη μύτη μα συμβαίνουν μπροστά, μα. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ελέγχουμε. Ευχαριστώ, Αγιούζο, και μετά, Γκίρλινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Αγιούζο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μα. Λοιπόν, μα είπε η ΕΦΣΑ ότι ε, δεν ε, έχει έγκυρη μεθοδολογία και απλώς ενδείξεις έχει για ενδεχόμενο κίνδυνο. Και μάλιστα αναθεωρεί αυτό τον καιρό τη μέθοδο αξιολόγησης κινδύνου. Ναι, δεν μας έκανα καμία σύσταση, ωστόσο εσείς ε, πήρατε την απόφαση να αποσύρετε αυτά τα προϊόντα για δύο χρόνια επειδή υπέγραψαν 75 βουλευτές ή τη 10% του κοινοβουλίου. Δεν ξέρω μήπως είδατε και από ποιες πολιτικές ομάδες ήταν αυτοί οι 75. Με εκπλήσει όσο και με ανησυχεί βαθύτατα η ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στην πίεση από κάποια μέσα ενημέρωση συγκεκριμένα και ε, δέχεται τις απαιτήσει τους χωρίς ε, βάσιμα επιστημονικά στοιχεία. Και σας ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το μέτρο στη Γεωργία διότι καμιά φορά παίρνετε μέτρα ε, για απειρή και μετά δεν κάνετε καμία αξιολόγηση. Για το κρέας του ύπου εγώ ανησυχώ Γιατί γίνονται αναλύσεις, διότι αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν απάτη ε, ως προς την ετικέτα, αλλά αυτό είναι και θέμα τη Επιτροπή Περιβάλλοντος, δεν θέλω να επιμείνω. Γκέρλινγκ και μετά Ράιμερς. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, μπορώ, έχω δύο ερωτήσεις. Ανησυχώ πάρα πολύ για τα νοικοτινοειδή Εσείς τι ε, ακριβώς ενιστάτε τώρα, γιατί έχει αλλάξει η σύσταση. Και τι γίνεται με το Βόλιο Κρέας έχει γίνει ενημέρωση στα κράτη-μέλη. Το 2009 άρχισε αυτή η ιστορία και δεν έχω βρει στοιχεία. Εκεί που εφαρμόζονται διάφορες απαγορεύσεις ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία και πριν προβείτε σε δρακόντια μέτρα μπορείτε να μας τα δώσετε για το κρέας που δεν έχω κανένα θέμα με τη δράση που αναλάβατε εσείς από τότε που ε, ξέσπασε το σκάνδαλο αλλά θέλω να μάθω για ποιο λόγο και σύμφωνα με τις δικές σας κατευθυντήριες γραμμές για το ε, θέμα από το χωράφι στο ράφι λέτε ότι έχετε ε, πει ότι την κύρια ευθύνη τη φέρουν τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνουν και τους ανάλογους ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετά και θα ελέγχει τις επιδόσεις των κρατών μελών με ε, έλεγχο ε, και επιθεώρηση. Δεν ρωτάω τι έγινε τον τελευταίο μήνα, ε, αλλά μήπως αυτά έπρεπε να είχαν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Η Μπρίτα Ράιμερς και μετά Τότς. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα κύριε Επίτροπε. Σύντομη ερώτηση για το ήπιο κρέας. Ε, επιτέλους καλό είναι που πήρατε μέτρα και ευχαριστώ την Ιρλανδία που αποκάλυψε αυτό το σκάνδαλο. Έρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Έχουμε αρκετή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τέτοιου είδους ελέγχους και μέτρα. Και δεύτερον, θα μπορούσατε ενδεχομένω να μας δώσετε μια επισκόπηση τις ε, δυνατότητες των εργαστηρίων των κρατών μέλων. Είναι αρκετά εξοπλισμένα, έχετε μια τέτοια αξιολόγηση. Για τη δέσμη των μέτρων για την υγεία πρέπει να πω ότι το θεωρώ καλό που επιτέλους ε, δρομολογείται και έχω και την περιέργεια να δω αν θα είναι πραγματικά απλούστευση. Θα το ε, λέξουμε πάρα πολύ. Και χαίρομαι αυτά που είπατε για τις ίες και για τις οτόχες όρνηθες. Ε, αφορά και τη δική μου χώρα, γιατί αυτό με τις χειρομητέρες δεν το τηρεί η Γερμανία, αλλιώς ε, γίνονται ε, στρεβλώσεις στον αγωνισμό και για τα novel food, το νέα τρόφιμα. Τελικά είναι πραγματικά επικίνδυνο για την υγεία του καταναλτού ένα κρέας αποκλωνοποιημένο ζώο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πολύ σύντομα, Επίτροπε, πρόκειται για θέμα απάτης, εγκληματικότητας. Ε, οι καταναλωτές αγοράζουν καλή την πίστη και έχουν εξαπατηθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν εδώ κάποια θέματα για τα οποία θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Ε, κάποιοι ήδη αναφέρθηκαν σε αυτά. Ε, το, το μήκος και οι περιπλοκές στην αλυσίδα τροφίμων. Θα πρέπει να τις συντομεύσουμε εάν προσέξουμε την ανιχνευσιμότητα στην περίπτωση αυτή. Είναι πολύπλοκη ε, διαδικασία και πώς θα επιβάλλει το νόμο τελικά η Υπηρεσία Ασφάλειας τροφίμων και πώς θα παρακολουθήσει την εφαρμογή. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της αξίας εντός της αλυσίδας τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε μια σειρά διευθυντών σούπερ μάρκετ που στην τηλεόραση είπαν «Συγγνώμη, εγώ δεν έκανα τίποτα, οι προμηθευτές μας τα κάναν όλα». Ε, έτσι μάθαμε ότι τα σούπερ μάρκετ πολύ λίγο ελέγχουν τα προϊόντα τους και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη θέση σας πάνω στο θέμα αυτό. πολύ σύντομα ε, δεν είναι γελίο το ότι η γεωργία στη χώρα μου μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική όσον αφορά την παραγωγή και ότι θέλετε, ε, ε, ε, μιλάτε για την απαγόρευση του των απαγορευμένων αυτών προϊόντων. Σμιτ και μετά Άντερσον. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. καταλαβαίνω, σε συμπονώ που πρέπει να απαντήσετε σε τόσες ερωτήσεις, αλλά και εγώ θα θέσω ερωτήσεις. Άκουσα αυτά που υπόθηκαν για την υπηρεσία προτύπων του, των τροφίμων και ο μόνος λόγος που προέκυψε αυτό το σκάνδαλο ήταν λόγω τυχαίου δειγματοληπτικού τεστ DNA ε, σε ένα κράτος μέλος. Ε, ε, κατά πόσο προτίθεστε να επεκτείνετε τις δοκιμές αυτές σε όλη την αλυσίδα τροφίμων και αναφέρομαι και στις ζωοτροφές, διότι φοβάμαι ότι θα δούμε πολλές εκπλήξεις όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Ω νομικό και ξέρω ότι είστε κι εσείς, ε, μου φαίνεται εκπληκτικό το, το ότι δεν ακούσαμε ε, για δίωξη ε, σε περίπτωση παραβίασης της σύμβαση ανάμεσα στον λιανοπολιτή και τον καταναλωτή, διότι το, και, το θέμα που τίθεται εδώ δεν είναι ο κίνδυνο για τον καταναλωτή, αλλά γνωρίζοντα το οι εξαμελίε έχουν παραπλανήσει τον καταναλωτή. Γνωρίζω ότι δεν είναι ακριβώ εντολή σα αυτό, δεν είναι ακριβώ αρμοδιότητά σα αυτό, αλλά σχετίζεται με τι αρμοδιότητέ σα. Ε, Μήπω λοιπόν θα πρέπει οι λιανοπολιτέ να φέρουν ε, ευθύνη. Ε, διότι ε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτά που λέγανε ότι δεν φταίνε οι ίδιοι. Σας παρακαλώ, έχουμε 12 εγγεγραμμένους και πρέπει να κλείσουμε σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα μερικοί να αποποιηθούν. Σας, θα σας αναφέρω τα ονόματα τώρα. Θα ήθελα μερικοί όμως να αποσύρουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε το σύστημα ευρωπαϊκής ε, ανιχνευσιμότητας είναι το πιο προηγμένο. Όμως τα συστήματα αυτά δεν ε, είναι ε, απόλυτα στοχοθετημένα, γι' αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο υπάρχουν μεγάλα κέρδη με μικρούς ε, κινδύνους και δεν υπάρχει επιμερισμός ευθύνης. Αυτό οδήγησε στο, ότι, στο να μειωθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή και πιστεύω ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και το θέμα της προέλευσης ε, και εδώ μιλώ για τα μεταποιημένα νοπά κρέατα ή τα κατεψυγμένα. Έτσι, τα κράτη θα είναι πλέον υπεύθυνα ως προς την αλυσίδα ε, προμηθειών και τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να είναι υπόλογα για το κρέας που πολλούν. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Επίτροπε τι, θα, ε, τι προτίθεστε να κάνετε ως προσλήψη συγκεκριμένων ε, μέτρων γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή νομοθεσία για τα ε, μεταποιημένα προϊόντα και τα κατεψυγμένα. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. Κόστιντζερ και Κορέια μετά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε. Ε, λέτε για το σκάνδαλο με το κρέας ύπου ότι ε, είναι θέμα σήμανσης και των κρατών μελών. Μα δεν επικρίνουμε εμείς την εσωτερική αγορά. Εμείς θέλουμε ο καταναλωτής να ξέρει τι αγοράζει, να γνωρίζει. Και διαφωνώ και με αυτό που λέτε ότι υπάρχει ε, σήμανση ε, χωρίς παραθυράκια και δεν έχει καμία σχέση. Μα ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει από πού προέρχεται ε, αυτό που τρώει και για το κρέας συγκεκριμένα πρέπει να ξέρει και που έχει εκτραφεί το ζώο και που έχει παραχθεί στη συνέχεια το τρόφιμο. Ακούμε συνέχεια ότι η βιομηχανία και το εμπόριο δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτό το κόστος. Μα στην Γεωργία όλο και περισσότερο εφευρίσκεται ε, διάφορα νέα ζητήματα και θα πρέπει να τα επομίζεται ο Γεωργός. Ε, με σήμανση, με έλεγχο, με δήλωση, αλλά αυτή τη στιγμή φεύγει από την εκμετάλλευση, ουδής πλέον σκοτίζεται για να το πω έτσι, ε, τι θα γίνει με το κρέας αυτό. Έχει έρθει η ώρα να ξαναδούμε τα θέματα της σήμανσης και να τα εφαρμόσουμε σωστά. Ε, ένα θέμα για τις ε, ΣΥΕΣ και την ομαδική, τον ομαδικό τους ενσταυλισμό. Είδαμε ότι έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές αυγών σε σκόνη ε, στην βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, ενώ η δική μας πτυνοτροφία πλήττεται. Για τα νέο νοικοτινοειδή η μελέτη από ό,τι είδαμε έχει λήψεις μπορείτε να αποκλείσετε και να δηλώσετε εδώ ότι δεν είναι το παραθεράκι για να μπουν οι μεταλλαγμένα στην Ευρώπη. Πρέπει να σας διακόψω. Στο τελευταίους δεν μπορώ να δώσω το λόγο ε, Κορέιτ και Ντελάνγκ. Διαδικαστικό. Ε, προβλέπεται έκτακτη συνάντηση Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 28 Φεβρουαρίου όπου ο Επίτροπος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα συνάδελφοι, ε, κάτι που δεν μπορεί να γίνει, να βρεθείτε σε αυτήν την έκτακτη, έκτακτη συνάντηση. Κορέα, καταρχήν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσία του. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με την, ε, να ασχοληθώ με την οδηγία περί καπνού. Η υγεία είναι πρώτη στο μέλημά μας, αλλά η νέα οδηγία αποτελεί ε, πνίγμα στην ευρωπαϊκή ε, καπνοβιομηχανία, διότι υπάρχουν νέες απαιτήσεις σε σχέση με την εμφάνιση αυτού του προϊόντος. Αυτό θα μπορούσε να πλήξει άμεσα ε, πολλές εκτάσεις καλλιέργειας καπνού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, κατά πόσο έχετε διενεργήσει μελέτες για τις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας που αφορά την Εστρεμαδούρα εύνη στην Ισπανία, όπου δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες εναλλακτικής ε, καλλιέργειας. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η Επιτροπή θα ε, προβλέψει νέες κατεξουσιοδότηση πράξης, έτσι ώστε να υπάρξει νέα, μια αναδιατύπωση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ε, θέλετε να εξετάσετε το θέμα των θερμοκηπίων όσον αφορά τις μέλισσες. Ε, περίμενα να μ' ακούσει ο Επίτροπος. Ε, όσον αφορά το αλογίσιο κρέας, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν μπορείτε να μα υποβάλλετε έκθεση σχετικά με τι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τι κυρώσει, διότι αυτή είναι η χιλιοστέρνα της Ευρώπης. Έχετε δίκιο. Δεν πρόκειται για έλλειψη νομοθεσίας, πρόκειται για έλλειψη ελέγχου και επιβολής των νόμων και επιβολής κυρώσεων. όσον αφορά τις, ε, μεταφορές, ε, τις οδικές μεταφορές, ε, έχει υποβάλει η Κομισιόν έκθεση σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να δω τις διαφορές στα κράτη-μέλη και στο θέμα αυτό. Κύριε Επίτροπε, θα βοηθήσει αν διαθέσουμε περισσότερα χρήματα στο Γραφείο Τροφίμων και κτηνιατρικής ε, ώστε να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και τέλος παρακαλώ να μας ε, δώσετε μια επισκόπηση σχετικά με το κρέας, ε, τα άλογα και το εμπόριο αυτών εντός της Ευρώπης. Τι δρόμους ακολουθούν. Πόλσον και Νταντέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είχα πάρα πολλές ερωτήσεις που θέλω να θέσω, αλλά δυστυχώς δεν έχω χρόνο όσον αφορά την επισήμανση και τον έλεγχο. Γίνονται ε, ε, ε, έλεγχοι DNA, τεστ DNA στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δοκιμές σε DNA στα τρόφιμα ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πολύπλοκη αλυσίδα τροφίμων. Και ε, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με το λογίσιο κρέας. Από πού προέρχονται όλα τα άλογα, ε, πώς μεταφέρονται και πώς ε, σφάζονται. Και αυτή είναι μια ερώτηση που μου θέτουν συχνά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μία παρατήρηση και μία πρόταση. Αυτή η ιστορία, το σκάνδαλο με το κρέας του αλόγου αποκάλυψε στο κοινό πόσο μακριά είναι η τροφική αλυσίδα ε, και η αγροτροφική. Το κοινοβούλιο έκανε μία πρόταση για την αλλαγή της λειτουργίας. Αφορά τέσσερις επιτρόπους αυτό. Έπρεπε το Δεκέμβρη να μας την είχατε καταθέσει. Τελειώνει ο Φλεβάρης, βγαίνει και ακόμα δεν μας την έχετε φέρει. Νομίζω αυτή η επικαιρότητα θα πρέπει να κινήσει λίγο τις εργασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μακρά λυσίδα λοιπόν και πού είναι η χνηλασιμότητα. Όταν είναι 4-5 οι φορείς θα πρέπει να είναι ε, υποχρεωτική έλεγχη για να είμαστε σίγουροι ότι έχει μέσα αυτό που γράφει η ετικέτα. Και όλα τα προϊόντα ε, που είναι εκτός προδιαγραφών και προτύπων είναι καλά προϊόντα και οι τράπεζες ε, τροφίμων ζητούν παρέκκληση για να δοθούν σε αυτές αντί να πεταχθούν τα προϊόντα. Παρακαλώ αυτά τα προϊόντα που έχουν κατασκευθεί να διατεθούν στις τράπεζες τροφίμων στην Ευρώπη γιατί έχουν μεγάλη ανάγκη λόγω και της κρίσης που ζούμε. Ε, Χόφμαν και μετά πατραωνέβεις; Μία λέξη θα πω για το Novel Food Deal. Ε, συμμετείχα σε ένα τριμερή διάλογο ο οποίος απέτυχε. Ελπίζω στο Novel Food να μην συμβεί κάτι παρόμοιο αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το Συμβούλιο. Στην αρχή συμφωνούσαμε, αλλά αποτύχαμε στην κλωνοποίηση μόνο. Όμως το κρέας ε, κλωνοποιημένων ζώων δεν θα μπει στη διατροφική αλυσίδα. Αυτό ε, το συμφωνήσαμε και ως προς το F1 είχαμε ε, συμφωνήσει ως προς την προέλευση από κλωνοποιημένα ζώα. Το ζήτημα αφορά τις κατηγορίες F2 και μετά. Είναι δύσκολη η ανιχνευσιμότητα σε αυτή την περίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στις ίδιες ε, ανησυχίες, λέει η κυρία Νέβες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το σκάνδαλο του κρέατος ε, αλόγου πλήττει ε, άλλους παραγωγούς κρέατος, ιδιαίτερα όταν το κρέας είναι από προέλευση αγελάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαταστήσουμε την εμπίστοσύνη του καταναλωτή. Το θέμα της ασφάλειας της διατροφικής αλυσίδας είναι ύψης της σημασίας, αλλά ο καταναλωτής θέλει και καινοτομία στα προϊόντα αυτά. Θα ήθελα να μας πει ο Επίτροπος τι πιστεύει γι' αυτό, γιατί δεν μας μίλησε για μελλοντικά σχέδια της Επιτροπής έτσι ώστε να προωθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, τις οποίες έχει εμπιστοσύνη ο κατανοητής Γκλάντενφέλντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε ότι θέλετε να περιορίσετε μόνο τη χρήση των νέων νοικοτινοειδών ε, στις περιπτώσεις που είναι απολύτως απαραίτητα. Ξέρετε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί είναι και πολλές ε, ε, διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν. Το είπα και προηγουμένω. Έχουν γίνει κάποιοι περιορισμοί πλέον στη χρήση αυτών των προϊόντων και για παράδειγμα οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι συνεργάζονται σε κάποιες χώρες όπως είναι η Ουγγαρία, η χώρα μου. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει δηλητηριαστεί καμία μέλισσα ε, από αυτές τις ουσίε. Αντίθετα, ε, όταν χρησιμοποιούνται τα υποκατάστατα, αυτά που μα προβάλλετε εσεί ω εναλλακτική λύση είναι ολέθρια και ε, οδηγούν σε μαζική εξαφάνιση ή αφανισμό των μελισσών. Θα ήταν λοιπόν η απαγόρευση στην Ουγγαρία πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μέλισσες, αν γυρίσουμε στα παλιά προϊόντα, να χρησιμοποιούνται σωστά και με μέτρο τα νέο νοικοτινοειδή. Και τα κράτη-μέλη δεν έχουν όλα τις ίδιες συνθήκες, ούτε το κλίμα, ούτε τα ίδια έντομα. Ο σκαραβαίος που πλήττει το καλαμπόκι μόνο με μεταλλαγμένα ή νεονικοτινοειδή ε, καταπολεμείται. Αυτά. Ε, επιτρέψτε λίγο στα κρατημέλη να δρουν ε, με κάποια ευελιξία. Ο Ερικ. Euh, Πρόεδρε, σε σχέση με το κρέας αλόγου θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για απάτη στην σήμανση, γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένους αδιφάγους προμηθευτές, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την διατροφική αλυσίδα με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν 750 ε, τόνοι κρέατος χιλιάδες τόνοι ε, να διακυβεύσουν το μέλλον της αγοράς. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες ανιχνευσιμότητας και σήμανσης καθώς και έλεγχη σε όλα τα κράτη-μέλη και να συντονιστούν οι έρευνες έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια ατυχή συμβάντα στο μέλλον. Οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ε, ε, μνήμα της προέλευσης του κρέατος και να ε, μιλάμε και για χρήση κρεαταλεύρων εκεί που γίνεται. Διαφορετικά θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ευχαριστώ συνάδελφοι. λυπάμαι κύριε Πίτροπε για, αυτό το, για αυτή τη χιονοστιβάδα ερωτήσεων, αλλά το θέμα, όλα τα θέματα είναι αρκετά επίκαιρα και πολλοί βουλευτές ήρθαν για να μιλήσουν από άλλες επιτροπές. Ελπίζω σε αυτά τα λίγα λεπτά να μας απαντήσετε κατά το δυνατόν. Ζητώ συγνώμη από τους διερμηνείς διότι έχει παραέλθει ο χρόνος. Μπορς. θα επιτύχω το αδύνατο, θα προσπαθήσω να επιτύχω το αδύνατο. Ας αρχίσω με το κρέας αλόγου και θα ήθελα να διασαφηνίσω κάτι. Γιατί μας εκπλήσει το γεγονός ότι αυτό το ανακάλυψε ένα κράτος μας, Δηλαδή ποιος άλλος θα έπρεπε να το ανακαλύψει. Τα κράτη-μέλη εγκρίνουν τα μέτρα, θέσεως σε ισχύ και δίνουν συνέχεια. Και η αντίδραση της Επιτροπής ήταν τάχιστη, γιατί όταν είδαμε ότι δεν ε, πρόκειται για μία ε, σποραδική, μία τυχαία περίπτωση μόνο στην Ιρλανδία και όταν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία και στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο, τότε η ανιχνευσιμότητα ε, ε, τέθη αμέσως ε, ισχύει το θέμα άρχισε από τη Ρουμανία, βγήκε το κρέας από τη Ρουμανία, πήγε στην Ολλανδία, μετά μεταποιήθηκε από μια γαλλική επιχείρηση στο Λουξεμβούργο και μετά διοχετεύθηκε στην αγορά από την μπίφλα λαζάνια. Δηλαδή, ο μηχανισμός ανιχνευσιμότητας ετέθη σε εφαρμογή άμεσα. Οι έρευνες δεν έγιναν αμέσως από τα κράτη-μέλη με αμεσότητα δηλαδή, αλλά όταν ήρθαμε σε επαφή με τα έξι κράτη-μέλη υπό Ιρλανδική Προεδρία, τότε ε, το κοινοποιήσαμε το θέμα και στη Europol, που δεν έχει το προσωπικό για τη διερεύνηση, αλλά χρειάστηκε να συντονίσει τις, δια... τις διαδικασίες διερεύνησης και ανακρίσεων στα κράτη-μέλη. Φυτεύω για δυόμιση μήνες, αλλά μπορώ να πω ότι δράσαμε τάχιστα. Στις 13 Φεβρουαρίου ε, συνήλθαμε με τα έξι κράτη-μέλη όπου εμφανίστηκε αυτό το θέμα. Έξι μέρες αργότερα βρεθήκαμε ενώπιον της ε, μόνιμης επιτροπής Εσείς μιλήσατε για μετριοπαθή σχέδια εποπτείας, όμως εγκρίθηκαν αυτά τα σχέδια εποπτείας και ελέγχου και μετά, δύο μέρες αργότερα, εγκρίθηκαν και στις 25 ε, Φεβρουαρίου θα το συζητήσουμε και στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που δεν ήταν θέμα διατροφικής ασφάλειας και το τονίζω για πολλοστή φορά. Αυτό είναι λανθασμένο. Εάν ήταν θέμα διατροφικής ασφάλειας, τότε θα είχαμε εγκρίνει τους συνήθεις κανόνες, δηλαδή να αποσύρουμε και να απαγορεύσουμε ορισμένα προϊόντα, διότι είναι επιζήμια για την ασφάλεια. Υπό τη ΣΑΝΚΟ υπάρχει και η επίσημη κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία δεν προβαίνει σε επιθεωρήσεις κρέατος ή υποπροϊόντων του, αλλά είναι θεματοφύλακας των θεματοφυλάκων, θεματοφυλάκων δηλαδή επιθεωρεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των κρατών μελών. Υπάρχουν 110 επιθεωρητές, οι οποίοι διενέργησαν 160-170 ελέγχους με αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα διατροφικής ασφάλειας και 75 σε τρίτες χώρες από όπου εισάγουμε κρέας και 13 ελέγχους στις χώρες υπό ενταξιακή διαδικασία αλλά δεν είναι εφικτό στο εγγύς μέλλον να έχουμε ένα σώμα επιθεωρητών που θα μπορούσαν in situ να δουν κατά πόσο η σήμανση είναι σωστή παντού. Θεωρητικά είναι δυνατόν, αλλά έμπρακτα αδύνατον υπό τις τρέχουσες συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας. Ακόμα και σε άλλα ε, θέματα ή χαρτοφυλάκια. Τι έχουμε, έχουμε ε, αρχές επιθεώρησης, ε, αρχές υπερεποπτείας δηλαδή, όχι επιθεωρητές που μεταβαίνουν επιτόπου για να ελέγξουν. Δεν υποβαθμίζω το γεγονός, αλλά ας αποδώσουμε ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. και ας εκτιμήσουμε τις προσπάθειες που καταβάλουν τα κράτη-μέλη στην ανείχνευση αυτών των παραβιάσεων στη διαδικασία σήμανσης και θα γίνουν οι κατάλληλες προσφυγές. Δηλαδή θα δούμε κατά πόσο χρειάζεται να εκκινηθεί μια ε, ποινική καθαρά διαδικασία. Τα σούπερ μάρκετ δεν είναι υπεύθυνα για λανθασμένη απατηλή σήμανση, αλλά οι προμηθευτές. Directive was also uh, mentioned and its effect. Και αναφέρθηκαν και οι επιπτώσεις ε, στις θέσεις εργασίας. Είχα παρόμοια ε, ερώτηση χθες στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και την επόμενη εβδομάδα ε, θα συζητήσουμε το θέμα της οδηγίας καπνού και είναι θέμα δημόσιας υγείας. Ε, η συνθήκη λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Η οδηγία αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των καπνιστών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελπίζω. Διότι, εάν όχι, δεν θα είναι αποτελεσματική. Εάν είναι αποτελεσματική, θα έχει οικονομικές συνέπειες εάν ε, μειωθεί ο αριθμός των καπνιστών ε, και αυτός είναι ο στόχος μας κατά 2% τα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρχουν οικονομικές συνέπειες. Ελπίζω να μην προτείνει κανεί ε, να προωθήσουμε το κάπνισμα για να δημιουργήσουμε περισσότερε θέσει εργασία στον τομέα του καπνού. Είναι λοιπόν κυρίω θέμα δημόσια υγεία. Θα υπάρχουν και οικονομικά πλεονεκτήματα ως αποτέλεσμα της οδηγίας που προτείνεται, διότι αν έχουμε μείωση των καπνιστών θα ε, εξοικονομήσουν χρήματα ε, από τον τομέα της υγείας ε, οι κυβερνήσεις, αλλά και ο πρώην καπνιστής τα χρήματα που θα εξοικονομήσει θα τα χρησιμοποιήσει σε άλλους τομείς της οικονομίας. Και ο στόχος της οδηγίας καπνού είναι να εναρμονίσει το μέγεθος ε, και την εμφάνιση των ε, πακέτων ε, τσιγάρων. Δεν θα πρέπει να μοιάζει με συσκευασία γλυκών, καραμελών ή αρώματος. Θα πρέπει να φαίνεται ότι είναι τσιγάρα και δεν προτείνουμε και και προτείνουμε ε, ενιαία ε, εμφάνιση. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι έχουμε ε, προχωρήσει υπερβολικά. Εγώ νόμιζω ότι αυτό ακριβώς δείχνει πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι αυτή είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση του θέματος. Προτείνουμε δηλαδή η συσκευασία να καλύπτεται από προειδοποίηση για την υγεία και μόνο το να αναγράφεται το όνομα της μάρκας. Πάντως νομίζω ότι είναι καλή η προσέγγιση αυτή. Επίσης, Θέλουμε το, ο καπνός να γίνει λιγότερο ελκυστικός. Δεν κρύβουμε την πρόθεση της Επιτροπής. Ε, η πρόθεσή μας είναι να μειώσουμε το κάπνισμα και τον αριθμό των καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το νεονικοτινοειδή, το θέμα δεν είναι να εξυπηρετούμε απλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να αντιδρούμε σε αυτά που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, στο θέμα αυτό. Ε, αντιδρούμε σε αυτά που μας λέει η ΕΦΣΑ. Η ΕΦΣΑ έχει εκπονήσει μια μελέτη η οποία κατέληξε ότι κάποια από τα νέα νοικοτινοειδή είναι βλαβερά για την υγεία των μελισσών. Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει ο Επίτροπος, θα πρέπει να αγνοήσει τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να απαντήσω στην Επιτροπή σας γιατί δεν ανέλαβα δράση δεδομένων αυτών που μας είπε η ΕΦΣΑ. Έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ. Επίτροπε, συγγνώμη πρέπει να σας διακόψω, θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, οι διερμηνείς πρέπει να αποχωρήσουν. Καλό σας βράδυ